Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο για την πέμπτη αυτή συνάντηση που οργανώνεται στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά που αισθάνομαι Το έχω τη δυνατότητα να κηρύξω την άναρξη αυτών των δύο ημερίδων εργασία. Και μάλιστα στη συνεργασία με τον συνάδελφο από την Τσεχική Γερουσία είμαι σε θέση να καλωσορίσω περί τους 100 εθνικούς βουλευτές. Και μάλιστα με εκπροσώπους από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την συμμετοχή σας σε αυτές τις ανταλλαγές απόψεων. Πριν προχωρήσω στις θέσεις που έχω να σας ε, απευθύνω ως προς τα δεδομένα που αντιμετωπίζουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και εσείς στα εθνικά σας κοινοβούλια, θα ήθελα να δώσω κάποιες τεχνικού χαρακτήρα πληροφορίες. Να σας υπενθυμίσω καταρχάς το πρόγραμμα ότι έχουμε δύο ημέρες εργασίας. Σήμερα με τον Επίτροπο Αλμούνια καταρχάς για θέματα μεταρρυθμισ... διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και βέβαια και με βάση το ερωτηματολόγιο που σας έχουμε υποβάλει θα προσπαθήσουμε, στόχος τουλάχιστον αυτό είναι, να ε, καταλάβουμε πώς μπορεί ο καθένας με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών να βοηθήσει τους υπόλοιπους ώστε να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις μεγάλες αυτές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και επίσης με την ανάπτυξη και εφαρμογή βέβαια των προγραμμάτων ανάκαμψης ίσως ο καθένας από το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο μπορεί να δώσει την ιδέα του για την δυνατότητα του Εθνικό Αυτό ε, να αναμειχθεί σε αυτό το σχέδιο ανάκαμψης και πάνω απ' όλα την υλοποίησή της. Στη συνέχεια θα έρθει και ο πρόεδρος Φιλίπ Μέιστατ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έναντι της οποίας ε, πολλοί απέναντι μάλλον στην οποία πολλοί ε, αναπτύσσουν τις ελπίδες τους, στρέφουν τα βλέμματα, περιμένοντας πρωτότυπες λύσεις και ε, προτάσεις για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων και δυνατότητες χρηματοδότησης για τις μικροπιστώσεις, δυνατότητες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η συζήτηση. Σήμερα θα έχουμε και συζήτηση με αξιωματούχο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου διότι δυστυχώ ο κύριο Μπούτρος Μπούτρο Γάλλη έχει ε, μείνει αποκλεισμένο στην Κουάλα Λουμπούρ και δεν υπάρχει δυνατότητα λόγω των αποστάσεων και των πτήσεων να έρθει σήμερα κοντά μα. αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα πιστεύω και με την παρουσία των δύο επιτρόπων του Λάσλο Κόβατ, υπεύθυνου για τα θέματα της φορολογίας και της κυρίας Νέλη, Νέλη που είναι υπεύθυνη για τον ανταγωνισμό να δούμε αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν τόσο πολύ. Αύριο προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων με τον Τσέχο Υπουργό Οικονομικών, που είναι και επικεφαλής του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ, κύριο Καφάλτσεκ, και τον κύριο Αλάστρο Πιγκάνη, που είναι στην ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπεύθυνο για τα διεθνή ζητήματα και πάνω απ' όλα το λεγόμενο δεύτερο Bretton Woods. κύριο Μπινισμάκη και που ασφαλώς θα είναι σε θέση να σα δώσει κάποιε ιδέε ε, και προτάσει. Έχετε βέβαια στο, στο σφακέλου σας τον κατάλογο των συμμετεχόντων αλλά και δύο έγγραφα που σα καλώ να πάρετε μαζί σα, Φαίνονται ίσω όμοια μεταξύ του, όμω διαφέρουν ω προ το εξή. Στα έγγραφα αυτά έχουν συμπληθεί αναλύσει των εμπειρογνωμών στους οποίους εμεί απευθυνόμαστε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα μάκρο οικονομικά και χρηματοπιστωτικών αγορών. Και τους ε, υποβάλαμε το ερώτημα, σε αυτούς τους εμπειρογνωμόνους που τακτικά συνεργάζονται μαζί μας, τους ζητήσαμε λοιπόν να εξετάσουν και να αναλύσουν τις εκτιμήσεις που από ευρωπαϊκής αλλά πάνω απ' όλα ανεξάρτητη σκοπιά θα μπορούσε να αναπτύξει θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, δηλαδή όχι από την πλευρά των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, ω προ την αποτελεσματικότητα και βέβαια τη πτυχή των σχεδίων ανάκαμψη, αλλά και των σχεδίων για υποστήριξη με ιδρύματα. Αυτά είναι τα έγγραφα λοιπόν, δυστυχώ μόνο στην αγγλική γλώσσα, αλλά ασφαλώ κάθε εθνικό κοινοβούλιο θα έχει κάποιου που θα είναι σε θέση να τα διαβάσουν και να αντλήσουν τι απαραίτητε πληροφορίε. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα την παρουσίαση που έχω να κάνω εγώ ως προς τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον συνάδελφο από την Τσεχική Γερουσία και ο Επίτροπος ο Τρίτος για τη δική του ανάλυση. Αυτή η πέμπτη μερίδα για μένα, όπως το υπογράμμισα άλλωστε και νωρίτερα, ξεκινάει με συναισθήματα συγκίνησης, αφενός, διότι ορισμένοι τους αδέλφους στο τέλος αυτής της θητείας θα αποχωρήσουν, κλείνει η θητεία μας το Μάιο, αλλά ταυτόχρονα και συνέστηση ευθύνη λόγω της μεγάλης οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε και η οποία, από την έποψη τουλάχιστον της ιστορίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μάλλον και η σοβαρότερη στην ιστορία μας. Επανερχόμενοι λοιπόν στις πατρίδες μας βλέπουμε όλοι πιστεύω την αγωνία των πολιτών, που στρέφονται προς εμάς και περιμένουν να τους στηρίξουμε. Εσάς, τους, ευρωβουλε... τους εθνικούς βουλευτές, εμάς τους ευρωβουλευτές, περιμένουν από εμά να επεξεργαστούμε, να αναπτύξουμε και να επεξεργαστούμε από κοινού λύσεις. Η κρίση μπορεί να ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει μείνει αλόβητη καμία περιοχή του κόσμου ύστερα από 1,5 χρόνο από την εκκίνηση αυτής της κρίσης, παρά τις όποιες ε, προσπάθειες για αποκόλληση από το άρμα αυτό, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για αποκόλληση και θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις τόσο προς το βράχι πρόθεσμο, το μέσο πρόθεσμο αλλά και τον μάκρο πρόθεσμο ορίζοντα, λύσεις που δεν θα είναι μεταξύ τους αντιφατικές. Και πρέπει να αναπτύξουμε προσπάθειες έτσι ώστε αυτές οι, προσπά... αυτές οι δράσεις που αναλάβουμε να βέρουν εκ παραλίλου και όχι σε σύγκρουση μεταξύ τοπικού, περιφερειακού, εθνικού ή ευρωπαϊκού επίπεδου. Δεν μπορούμε να πούμε «Α, η κρίση είναι παγκόσμια, περιμένουμε να βρεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο μία λύση για να προχωρήσουμε εμείς σε ανάπτυξη δράσεως σε εθνικό επίπεδο». Όχι, στα τρία επίπεδα, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Αυτό είναι το καθήκον μας. Και οι μέρε αυτέ, όπω σα είπα, είναι και ευκαιρία για ανάπτυξη ενό απολογισμού οικονομικού και χρηματοπιστωτικού για την Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμω, και πέραν αυτού του απολογισμού, όπω έλεγα κοινότερα, θα πρέπει να αναλογιστούμε τα συλλογικά ε, τις συλλογικές θέσεις, συλλογικές απαντήσεις που μπορούμε να προσφέρουμε για την κρίση αυτή και ενδεχομένως να στήσουμε νέες λύσεις. Αντιμετωπίσουμε λοιπόν μια παγκόσμια κρίση που ξεκίνησε από την αποτυχία του συστήματος των subprimes που οδήγησε σε ε, καταρρεύσεις οικονομικές ε, που βλέπουμε να προκαλούν οδυνηρές συνέπειες σε κάθε χώρα. Πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε τη λειτουργία των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών μας πάνω από όλα συστημάτων και αυτό γρήγορα, αποτελεσματικά, στοχευμένα αλλά και κατά τρόπο συντονισμένο, συνεργατικό, εστιασμένο. Είναι βέβαια οι οικονομικές ε, και ε, δημοσιονομικές αρχές σε θέση και απαραίτητο να συνεργαστούν μεταξύ τους και μόνο με συντονισμό, συντονισμένη δράση μπορούμε να δώσουμε οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική λύση όπως τη χρειαζόμαστε. Η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγαρών και πάνω απ' όλα η εποπτεία αυτών δεν είναι κενά, κενά δηλαδή καινούρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήματα. Έχουμε επανειλημμένο ζητήσει την ε, την ενίσχυση της εποπτείας στις μοτοπιστωτικές αγορές. Άλλωστε ξέρετε ότι αυτό και πέρυσι μας είχε απασχολήσει ιδιαίτερος με την παρουσία στη συζήτησή μας του Βαρόνου Λαμφαλούση όπου επιμείναμε ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά. Με πρόσφατη έκθεσή μας εξάλλου πολύ συγκεκριμένα επενθυμίσαμε την ανάγκη για εποπτεία των δια ή υπερσυνοριακών ομίλων. Σήμερα και καθώς είναι τόσο κατεπίγουσα η ανάγκη για την ανέβρεση λύσεων, θα ήθελα και εγώ ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπογραμμίσω ότι έχουμε αρκετές προτάσεις ακούσει για τροποποίηση της υφιστάμενης χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Έχουμε την εντύπωση όμως και πρέπει να το ομολογήσω αυτό ότι η δουλειά του νομοθέτη ίσως πότε πότε να οδηγεί σε σοβαρή απογοήτευση διότι νομοθετούμε επί τη βάση μια αρχιτεκτονική, η οποία κινείται διαρκώ, μεταβάλλεται διαρκώ. τα νέα τη θεμέλια δεν έχουν προσδιοριστεί ή δεν έχουν πάντω παγιωθεί επαρκώ. και η προσέγγιση μερικέ φορέ είναι μόνο τομεακή και ίσω να φαίνεται και πεπαλαιωμένη. Μπορεί να είμαστε πολύ αποφασισμένοι σε δράση και σε έγκαιρη δράση, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη είναι αναγκασμένη πολλέ φορέ να ανοίξει τι αγορέ τη απέναντι στον ανταγωνισμό και να κυνηγάει Τρέχοντα από πίσω την καινοτομία διαφόρων παραγόντων των αγορών χωρί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη ρήξη της ισορροπίας που μπορεί μια τέτοια καινοτομία ή νέα συστήματα να, να προκαλέσει στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σήμερα αντιμετωπίζουμε σοβαρέ δυσκολίες δεινέ συνθήκες, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αρχιτέκτον να αναλάβει δράση το ταχύτερο δυνατό και να εκφράσει μέσα σε ευρωπαϊκό νομοθέτημα τις ρυθμίσεις που θα προκύψουν από τις προτάσεις και τις συζητήσει τη ομάδα που έχουν αναπτυχθεί ε, περί τον πρόεδρο Ζακ Ντελαγοζιέχ. Ζητούμε πολλά, αναμένουμε πολλά μάλλον από την ομάδα αυτή αναλογισμού για νέε σύγχρονε ευέλικτε λύσει για την κοινοτοπιστωτική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να παραμείνει αυτή και ανεξάρτητη ενεργειακά και να την ασυνθέσει να αντιμετωπίσει τι κλιματικέ αλλαγέ, αλλά και να διατηρήσει την κοινωνική τη συνοχή. Το σύστημα τη εποπτεία δεν θα πρέπει να αναζητήσει σε απίθανα μέρη τι εμπνεύσει του. Πιστεύουμε ότι ένα Ευρωπαίο επόπτη μπορεί να ακολουθήσει το σύστημα της εποπτείας των ε, κεντρικών τραπεζών, όπου ο καθένας ανεξαρτήτως των διαστάσεων της χρηματοπιστωτικής του αγοράς θα βρίσκει τη θέση του, θα αισθάνεται στα νερά του μέσα, θα μπορεί δηλαδή να συνδυάζει και τις γνώσεις του, αλλά και την ευρωπαϊκή δράση, αλλά και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Στο πλαίσιο αυτό ε, μπορούμε να έχουμε και τη διασύνδεση με την κεντρική τράπεζα στο πλαίσιο της μακρο και προληπτικής εποπτείας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ενισχυθεί από τη δοκιμασία αυτή και χάρη στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση. Με την επιδείνωση όμως της κατάστασης διαπιστώνουμε ότι οι παρεμβάσεις των κρατών κρίθηκαν απαραίτητες. Για το μέλλον θα πρέπει να αναλογιστούμε ποια θα είναι η δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρειαζόμαστε για το μέλλον και εγώ προσωπικώς θα ήθελα, αν το επιτρέπετε, να εκφράσω τη σκέψη ότι θα πρέπει ενδεχομένω να αναδιοργανωθούν κάποιε πτυχέ τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι μακροοικονομικέ πτυχέ, οι πτυχέ τη διαχείριση των, ε, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα έπρεπε ενδεχομένω να υπαχθούν σε μία υπηρεσία από κοινού για την ανάπτυξη, ανάκαμψη των οικονομικών προσπαθειών. Θα πρέπει να μην μείνει ω μοναδικό στόχο η μονομανία, η σταθεροποίηση τη ε, οικονομία. ή ο περιορισμός των ε, δαπανών των κρατών. Ο φάρος αυτός θα έλεγα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η απομόνωση ή ο απομονωτισμός είναι ο μεγάλος κίνδυνος που επαπειλείται και που μπορεί να μας οδηγήσει σε τεράστιους σε τεράστια σφάλματα. Βλέπουμε κάποιες τέτοιες παρεκκλήσεις μέσα στο ΕΚΟΦΗ να εκφράζονται όταν κάποια κράτη αρνούνται να αξιοποιήσουν το περιθώριο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ε, από τον προπολογισμό μόνο ε, για να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή προσπάθεια. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος διάρρηξης της ζώνης του ευρώ. Η έξοδος από ένα κράτος για ένα κράτος από τη ζώνη του ευρώ θα σημαίνει ακόμα δυνότερες συνθήκες και περιστάσεις. Δεν νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον ουδήποτε κράτος τη ζώνη ευρώ να αποχωρήσει ή να δεχθεί την αποχώρηση κάποιου άλλου. Η συνθήκη αποκλείει το λεγόμενο bailout, δηλαδή την αυτοεξαίρεση, αλλά πρέπει να επιδείξουμε και εφευρετικότητα, δημιουργικότητα για την, ε, στην αναζήτηση των λύσεων όπως χρειάζεται κράτη έξω από τη ζώνη, αλλά πολλές φορές και από την Ευρω... έξω και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, βλέπουν πλέον εκτίματα από την δυνατότητα της προσχώρησης. Πρέπει αυτό να το αξιοποιήσουμε. Δέκα χρόνια εορτάζουμε από την θέσπιση του ευρώ. Κάποια από τα κράτη σας μόλις εντάχθηκαν στο ευρώ. Κάποια άλλα προσπαθούν να μπουν στη ζώνη του ευρώ. Το ευρώ είναι επιτυχία και είμαστε υποχρεωμένοι να τη διατηρήσουμε και να την αναπτύξουμε περισσότερο. Οι αποκλήσει που εμφανίζονται στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ των κρατών μπορεί να μεγαλώσουν αν χάσουμε αυτό το μεγάλο ατού που είναι το ευρώ. Άλλωστε, επεσήμανε και στην πρόσφατη έκθεσή του, πριν από ένα περίπου χρόνο, ο ε, Επίτροπος Αλμούνια τους κινδύνους αυτούς. Εάν δεν συνεχίσουμε την προσπάθεια, αν δεν μεγεθύνουμε το ευρώ, κινδυνεύουμε, κινδυνεύουμε να χάσουμε και την ε, έννοια της εμπιστοσύνης στο σύμφωνο σταθερότητας, την ασφάλεια των αγορών και ως εκ τούτου πρέπει να αναπτυχθεί και μια νέα στρατηγική, μια στρατηγική που θα την ε, ε, ονόμαζα στρατηγική όλοι βγαίνουν κερδισμένοι και μια στρατηγική η οποία δείχνει ότι μπορούμε το 60% του ΑΕΠ μας να το αξιοποιήσουμε, να το χορηγήσουμε τρόπον κοιτινά σε ένα σύστημα αμοιβαίας εμπιστοσύνης αλλά και αμοιβαίας εποπτείας. Ένα σύστημα ενίσχυσης της λειτουργίας της Ευρωζώνης. Κάποιοι θεωρούν ότι οι αποκλείς μέσα σε μια ε, νομισματική ζώνη να μην έχουν πολύ μεγάλη σημασία και να παραπέμπουν επί στο παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών όπου όμως είναι μεγάλη διαφορά διότι το 3% του ΑΕΠ ανήκει στον ομόσπονδο ομοσπονδιακό καλύτερα προπολογισμό. Πράγμα που διαφέρει πολύ από τα ποσά τα οποία γνωρίζουμε εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτέ ήταν κάποιε ιδέε που πιστεύω τροφοδοτούν τη συζήτηση. Πεποίθησή μου είναι τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο καθένα διαρωτάται ποια θα είναι η δεύτερη, ε, το δεύτερο ρεύμα, το δεύτερο κύμα ε, κρατικών ενισχύσεων ή στηρίξεων ή καθένας διερωτάται τι μπορεί να προσφέρει ως λύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Σύνοδο Κορυφής των G20 και ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέλος σε αυτή την σύνοδο, κατά τη στιγμή κατά την οποία γίνεται η προετοιμασία και του έκτακτου Συμβουλίου Κορυφής, έχουμε πιστεύω μια εξαίρετη ευκαιρία και να ανταλλάξουμε ε, απόψεις ή να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας, αλλά πάνω απ' όλα να αναζητήσουμε λύσεις για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ και ας δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο από την Τσεχική Γερουσία για να ακούσουμε τις δικές του απόψεις. Κύριε Συμπρόεδρε, έχετε το λόγο. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Με μεγάλη μου χαρά αλλά και τιμή συμμετέχω σήμερα σε αυτή τη ε, συζήτηση για το μέλλον της οικονομίας της Ευρώπης και για άλλη μια φορά. Συναντιόμαστε αγαπητέ Πρόεδρε που συναντηθήκαμε τον Νοέμβριο πέρσι για πρώτη φορά τότε σε εκείνη την συνεδρίαση την ε, οικονομική με την ε, Επιτροπή ε, Γεωργίας και Μεταφορών στην οποία εγώ συμμετέχω θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε ε, προς μια οικονομική ανάπτυξη με επιτυχίες ταυτόχρονα και στα μέτωπα της ε, κερνοτομίας, της ε, έρευνας και των ΜΜΕ. Ξεκινάω από αυτό το τελευταίο το οποίο αναφέρθηκε, δηλαδή της ΜΜΕ και συμφωνώ με αυτά τα οποία άκουσα. Ξέρετε, αύριο θα έρθει ο Υπουργός Οικονομικών, θα σας μιλήσει για τις προτεραιότητές μας, για τα οικονομικά ζητήματα για πάρα πολλά θέματα, οπότε θα μπει στις λεπτομέρειες ε, και φαντάζομαι ότι εσείς θα συμφωνείτε ότι η ραχοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι η ΜΜΕ. Χρειάζεται ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αυτό είναι το κλειδί, ούτως ώστε να υπάρχει υγιές επιχειρηματικό κλίμα. Άρα χρειάζεται εύστοχη νομοθεσία, φιλική στις επιχειρήσεις. πολυνομία είναι ένα πρόβλημα. Και γι' αυτό βασική προτεραιότητα της Τσέχικης Προεδρίας είναι να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Το Δεκέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε ένα καινούριο πλαίσιο ε, για να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η Τσεχική Προεδρία πρόθεσε την υπόθεση αυτή η δε γερουσία της Τσεχίας επίσης νομοθέτησε για τις ΜΜΕ ε, και κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων την ένταξή μας. Οπότε θέλουμε να καταβληθεί πάσα δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε οι αρχές που περιέχονται στο νομοθέτημα εκείνο να είναι νομικά δεσμευτικές και επίσης ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογή αυτού του νομοθετήματος σε κοινοτικό επίπεδο, στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας, αλλά και σε επίπεδα εθνικά, στα πλαίσια των εθνικών ε, σχεδίων και προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να δούμε ποιες είναι οι πιο άμεσες λύσεις ε, Ποιε είναι οι πιο προβλημένες λύσεις. Πάντως θα, πρέπει να δούμε πιο μακρόπνο, να δούμε το ότι δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει η Ευρωπαϊκή Οικονομία. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε ευκαιρία να μιλήσω. Ευχαριστούμε Ευχαριστώ, εμείς κύριε... κύριε Πρόεδρε για αυτή την ε, πολύ σαφή προσέγγισή σας και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, επίτροπο ο οποίος είναι εδώ. Ξέρουμε όλοι ποιες είναι οι προσμονές και οι προσδοκίες οι οποίες υπάρχουν γύρω από το χαρτοφυλάκιό σας και σας δίνω το λόγο για να μπορέσετε να μας παρουσιάσετε την οικονομική κατάσταση και πώς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να συμβάλλει στη συζήτηση για τις μακροοικονομικές τους μακροοικονομικούς ε, προβληματισμούς που υπάρχουν. Ευχαριστώ κύριε κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Δεν μπορώ να μιλήσω στα καταλανικά για τον συνάδελφό μου και το συμπατριώτη μου. Πρώτα απ' όλα όμως όσον αφορά την οικονομική κατάσταση Έχουμε, είχαμε προβλέψει για ε, φέτος ε, μία πρόβλεψη την οποία θα παρουσιάζαμε κανονικά το Φεβρουάριο αλλά την παρουσιάσαμε ήδη στις 19 Ιανουαρίου δηλαδή πριν τρεις εβδομάδες και όπως άλλωστε έγινε και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις προβλέψεις του ΟΣΑ και τις προβλέψεις διαφόρων ιδιωτικών και δημοσίων οργάνων έχουμε προσαρμόσει πολύ ε, τα επίπεδα αναπτύξεως και ποσοστού απασχόλησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποχρεωθήκαμε να αυξήσουμε ή ε, να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω τις ε, προβλέψεις μας για τους αριθμούς ανεργίας για το τρέχον έτος στην, ε, οικονομική, στην ευρωπαϊκή οικονομία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σε όλη την Ευρώπη αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σε σοβαρή ύφαση, ύφεση όπως άλλωστε ισχύει για τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, την Ιαπωνία και άλλες οικονομίες διεθνώς και η ανάπτυξη για εφέτος θα προκληθεί από τις αναδυόμενες οικονομίες οι οποίες όμως επίσης χρειάστηκε να μειώσουν τις προβλέψεις τους για την Κίνα δηλαδή τουλάχιστον πέρυσι είχαν καταγράψει ένα ποσοστό ανάπτυξης 9, 10, 11% και φέτος σύμφωνα με τις προβλέψεις μας θα έχουν μια ανάπτυξη γύρω στο 6%. Υπάρχει λοιπόν μια ουσιαστική ε, αναθεώρηση προς τα κάτω ακόμη και για την Κίνα, για την Ινδία μια άλλη σημαντική αναδυόμενη οικονομία την ε, περασμένη εβδομάδα σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επισκεφθήκαμε τη Ρωσία και η ρωσική οικονομία έχει επίσης ε, σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε στο ότι ε, θα αντισταθμιστεί η έλλειψη εσωτερική ζητήσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως άλλωστε και στις Ηνωμένε Πολιτείε μέσω της εξωτερική ζητήσεως που θα προκληθεί από τις αναδυόμενες οικονομίες. Υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα, είναι η πρώτη ύφεση στην παγκόσμια οικονομία και είναι μια πολύ σοβαρή ύφεση. Τι αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε. Όπως θυμάστε, πρώτα απ' όλα αντιμετωπίσαμε μία οικονομική κρίση από τον Αύγουστο του 2007 και σε, Ευρωπα... Ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και συνολικά θελήσαμε να βελτιώσουμε τους οικονομικούς κανονισμούς, να συντονίσουμε καλύτερα την εποπτεία των τραπεζών, να επιλύσουμε τις ε, δυσλειτουργίες ε, των... του χρηματοοικονομικού συστήματος δεν είναι μόνο χρηματοοικονομική αλλά και οικονομική καθαρά κρίση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το φθινόπωρο να υιοθετήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανακάμψεως με οικονομικά κίνητρα για το 2009 και τα κίνητρα αυτά, τα φορολογικά, θα υιοθετηθούν σε εθνικό επίπεδο διότι οι προπολογισμοί ουσιαστικά είναι ακόμη εθνικοί και ε, ο συντονισμός είναι ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του προγράμματος ανακάμψεως γιατί τα κίνητρα θα είναι αποτελεσματικά εάν υπάρχει συντονισμός. Θα μπορούν να αποδώσουν αν όλες οι εθνικές αποφάσεις συντονιστούν επαρκώς και εάν το μέγεθος των φορολογικών κινήτρων μπορεί να συνδυαστεί με το χώρο ελιγμών που θα προσδώσουν αυτά τα φορολογικά κίνητρα στις εθνικές οικονομίες και αν από την πλευρά των εσόδων του προπολογισμού τα μέτρα θα είναι έγκαιρα, συγκεκριμένα και περιορισμένα χρονικά. Δηλαδή αυτή είναι η στόχη του προγράμματος μας ανακάμψεως το οποίο υιοθετήθηκε από τους 27 ε, αρχηγούς κρατών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Πολλές χώρες λοιπόν είχαν ήδη υιοθετήσει για τα φορολογικά κίνητρα προγράμματα τα οποία συνάδουν με ε, αυτό το προγραμματισμό σεισμό. Προχθές και ε, σήμερα μπορώ να σας πω προχθές στο Συμβούλιο και σήμερα εδώ μπορώ να σας πω ότι οι εθνικές αποφάσεις που ελήφθηκαν σχετικά με τα σχέδια εθνικής ανάκαμψης είναι ευθυγραμμισμένα με ε, τις ε, προβλέψεις που είχαμε δηλαδή περιορισμένου χρόνου συγκεκριμένα και εστιασμένα σε γενικές γραμμές τουλάχιστον συνάδουν με αυτές τις προϋποθέσεις για να υπάρξει μια αποτελεσματικότητα των φορολογικών ε, μέσων, μέτρων και όταν ε, συγκεντρώσουμε όλα τα εθνικά προγράμματα βλέπουμε ότι αντιπροσωπεύουν ε, περίπου 1% του ΑΕΠ δηλαδή λίγο λιγότερο από ό,τι είχε προβλεφτεί και συγχρόνως ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη έχει υπάρξει ένα άλλο είδους μέτρων το οποίο είχε υιοθετηθεί για να αυξηθεί η οικονομική στήριξη των οικονομιών και οι αυτόματοι σταθεροποιητές των ευρωπαϊκών οικονομιών λειτουργούν και πιστεύουμε ότι η επίπτωση των φορολογικών κινήτρων για την οικονομία για το τρέχον έτος το 2010 βάσει αυτών των μέτρων μπορεί να αξιολογηθεί σε 3,3 έως 4% του ΑΕΠ. Δηλαδή πρόκειται για ένα σημαντικό φορολογικό ε, κίνητρο όσον αφορά τις μεσοπτώθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές αυτών των δράσεων πρέπει να πούμε ότι ορισμένα μέτρα είναι στενά συνδεδεμένα με τις διαρθρωτικές αναθεωρήσεις οι οποίες χρειάζονται για να ενισχύσουμε τις οικονομίες μας και να ετοιμαστούμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα για μία σταθερή ανάκαμψη άπαξ και οικονομική κρίση και τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα επιληθούν και εξαφανιστούν. Υπάρχει λοιπόν μια καλή διασύνδεση μεταξύ των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί που θα φέρουν ε, βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική λαμβάνοντας υπόψη τις διορθωτικές ανάγκες ε, των οικονομιών μας. Συγχρόνως όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο περιορισμούς βραχυπρόθεσμα. Ο πρώτος περιορισμός είναι η κατάσταση των οικονομικών αγορών του τραπεζικού τομέα ιδίως και όχι μόνο του τραπεζικού τομέα αλλά και ορισμένων κεφαλαιοαγορών οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά και σε ορισμένες υπόψεις, περιπτώσεις δεν λειτουργούν καθόλου. Μαζί με τα φορολογικά κίνητρα τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν το τελευταίο τετράμινο πάρα πολλά προγράμματα, πρωτοβουλίες, έλαβαν αποφάσεις για να στηρίξουν τον χρηματοοικονομικό τομέα και να αποκαταστήσουν την ε, εύρυθμη λειτουργία των χρηματαγωγών μετά από την πτώχευση της Lehman Brothers 15 Σεπτεμβρίου όπου υπήρχε μια κατάρρευση του χρηματοοικονομικού συστήματος και αντιδράσεις των κεφαλαιογορών σε αυτή την κατάρρευση τα κράτη-μέλη είχαν υιοθετήσει ένα μακρύ κατάλογο μέτρων στηρίξεως ε, αναδιάρθρωση κεφαλαίου μεγαλύτερη ρευστότητα η οποία προσεφέρθη από τις κεντρικές τράπεζες ε, περικοπές των επιτοκίων και ούτω καθεξής και όλα αυτά τα μέτρα άρχισαν να επιδρούν θετικά σε ορισμένες περιπτώσεις ε, και στις κεφαλαιογορές μειώθηκαν οι διαφορές στο γιούρι και σε άλλα μέτρα από όταν υιοθετήθηκαν ε, αυτά τα κίνητρα αλλά εχθές συζητήσαμε στο επίπεδο του ΕΚΟΦΗΝ πώς ε, ε, θα λύσουμε το πρόβλημα του ενεργητικού το οποίο έχει εξαφανιστεί και αυτό ισχύει και επηρεάζει πολύ ορισμένα κράτη-μέλη και συγχρόνως λοιπόν θέλαμε ε, εφόσον έχουν, ε, έχει μειωθεί το ενεργητικό και έχει πληγεί ε, να προωθήσουμε νέα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να στηρίξουν το οικονομικό σύστημα και θα μπορέσουν να επαναφέρουν σε μία εύρυθμη λειτουργία των χρηματαγορών. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα από κοινού θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε μια θετική εξέλιξη των οικονομιών μας αλλά είμαστε βέβαιοι ότι αν οι χρηματαγορές και οι οικονομικές αγορές δεν λειτουργήσουν πιο εύρυθμα στους επόμενους μήνες η αποτελεσματικότητα των φορολογικών κινήτρων μας και της χρηματικής πολιτικής θα επηρεαστεί αρνητικά και σημαντικά. Και το δεύτερο θέμα στο οποίο ε, πρέπει να σταθούμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες είναι το γεγονός ότι δεδομένου του υψηλού ποσοστού δημοσίων πόρων που εμπλέκονται εις ε, τα οικονομικά κίνητρα και στα τα ε, χρηματοοικονομικά πακέτα έχει μεταφερθεί το βάρος από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο τομέα από τα ιδιωτικά κεφάλαια στα κρατικά κεφάλαια και ορισμένα κράτη-μέλη αρχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή επιπλέον δυσκολίες να χρηματοδοτήσουν το δάνειό τους και να εκδώσουν νέα ομόλογα για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις που έχουν λάβει αυξάνουν δηλαδή ε, τα χρέη τους και το κόστος της χρηματοδοτήσεως ε, των ε, χρεών στις περισσότερες χώρες αυξάνει διότι αυξάνονται και τα επιτυχία το δανεισμού όχι μόνο εις δημόσιες αγορές αλλά και στις ε, ιδιωτικές αγορές. Πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν όλα αυτά τα όρια και όλα τα κράτη δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες να αυξήσουν τα χρέη τους και να μπορέσουν να ε, χρημα το δοτήσουν τα κρατικά τους ομόλογα και ε, να διοχετεύσουν ρευστότητα στην αγορά τους. Αυτά είναι, λοιπόν, αυτές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μαζί με τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης και της σημαντικής επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας από πλευράς ανεργίας και καταστροφής θέσεων εργασίας. Γι' αυτό το λόγο οι συνεδριάσεις, οι διασκέψεις κορυφής, οι πρωτοβουλίες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ κατά τους τελευταίους μήνες. Και σήμερα έχουμε μία συνεδρίαση στο κτίριο του Μπερλεμό δηλαδή στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με ε, τον Πρωθυπουργό Πολάνικ και με τον Πρόεδρο Μπαρόζο μετά από τη συνάντησή τους στη συνέντευξη τύπου είπαν ότι μετά από τη διάσκεψη κορυφής που ανακοίνωσαν ε, εχθές ε, θα διοργανωθεί η συνάντηση στην 1η Μαρτίου και θα ε, υπάρξει στις 19 του Μαρτίου πάλι ε, ε, μία διάσκεψη των αρχηγών κρατών και προηγουμένως 22 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο μία συνάντηση των οικονομικών υπευθύνων και όλες αυτές οι συνεδριάσεις θα προετοιμάσουν τη συνάντηση των G20 στο Λονδίνο και ε, σήμερα οι κύριοι Τοπολάνη και Μπαρόζο είπαν ότι μια νέα διάσκεψη κορυφής θα γίνει στην Ευρώπη το Μάιο για να συζητήσουμε συγκεκριμένα την απασχόληση, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία και να βελτιώσουμε την κατάσταση των αγορών εργασίας. Αυτές είναι πολύ σημαντικές και πολύ ισχυρές ενδείξεις της ε, ε, υπάρξεως της Ευρώπης, της δυνατότητας να λύσει το πρόβλημα, να υπάρξουν κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μία κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο παγκόσμιο επίπεδο, είτε πρόκειται για τους G20 είτε παγκοσμίως. Και αυτά τα νέα είναι πολύ καλά νέα. Επίσης είναι πολύ καλό νέο διότι δίδεται το μήνυμα στους οικονομικούς παράγοντες και στους πολίτες ότι οι οικονομικοί θύνοντες γνωρίζουν το πρόβλημα αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητά του, αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις και έχουν αποφασίσει να τις αντιμετωπίσουν και να λύσουν τα προβλήματα άμεσα. Δεν μπορούμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις αυτές σε εθνικό επίπεδο μεμονωμένα αλλά με τους εταίρους της Ευρώπης θα πρέπει να τη και δεν μπορούμε να απομονωθούμε και από την παγκόσμια οικονομία. Θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να δώσει αυτές τις απαντήσεις. Τι απαντήσεις χρειάζονται. Αναλύσαμε με μεγάλη ανησυχία ορισμένες ενδείξεις εντός της Ευρώπης και εκτός της Ευρώπης ορισμένες ενδείξεις προστατευσισμού και πρέπει να είμαστε σαφείς. Σήμερα το πρωί ήμασταν σαφείς στις συζητήσεις μας όπως ήμασταν και χθε εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και έχουμε δεσμευτεί να προστατεύσουμε τους ανθρώπους ε, από τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσεως και να βοηθήσουμε τις κοινωνίες μας να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες το ταχύτερο δυνατόν θέλουμε να προστατεύσουμε τις οικονομίες μας, τους οικονομικούς τομείς, τους οικονομικούς παράγοντες, να τους δώσουμε τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση. Αλλά είμαστε κατά του προστατευτισμού και δεν είναι δυνατόν να θέσουμε στο ίδιο επίπεδο την προστασία των ατόμων και των οικονομικών παραγόνων δεν μπορούμε να τα ευθυγραμμίσουμε με προστατευσισμό. Αυτό είναι η χειρότερη λύση, η χειρότερη απάντηση σε αυτό το πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφώ. Εμεί ε, έχουμε δεσμευτεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι σίγουρο ότι αυτό αφορά και τα άλλα θεσμικά όργανα όπω και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και εθνικά θεσμικά όργανα των κρατών Όλοι έχουμε δεσμευτεί να προστατεύσουμε την εσωτερική μας αγορά και να καταπολεμήσουμε ουδίποτε είδου είδους φραγμούς, διακρίση μέσα στην εσωτερική αγορά και έτσι να είμαι ε, έτοιμοι να βρούμε κάποια απάντηση, κάποια απόκριση κοινή που να έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα. μια τέτοια κρίση θα πρέπει να εντοπιστεί με περισσότερη δράση πλευρά της Ευρώπης, όχι με λιγότερη. Και θα πρέπει να προστατεύσουμε όχι μόνο την εσωτερική αγορά, όχι μόνο τους ε, κανόνες του ανταγωνισμού. Αυτό είναι το, το, το ελάχιστο το οποίο απαιτείται. Ε, βέβαια, φυσικά και αυτό ισχύει τους, ε, τους καλούς καιρούς. Επίσης θα πρέπει κανείς να προστατεύσει το πιο σημαντικό αγαθό και μέσο που έχουμε στα χέρια μας, ε, αυτό το οποίο μας δίνει ένα όπλο κατά τη ύφεσης και να δούμε κατά πόσον είναι δυνατόν να έχουμε μια κοινή προσέγγιση σε αυτή την συγκυρία και έτσι να μπορούμε να έχουμε μια ε, νομισματική ε, ένωση. Μας προστατεύει το ευρώ. Μας δίνει ένα καταφύγιο, μια ασπίδα. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ θετικό ε, μέσο, τόσο ώστε να μπορέσουμε να χειριστούμε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, κρίση και όχι, όχι μόνο αυτούς τους 330 εκατομμύρια Ευρωπαίους και αυτά τα 16 ε, κράτη. Μιλούμε για όλους τους Ευρωπαίους. Όμως, ως Ευρωπαίοι και ως Ευρωπαϊκά Δεσμικά Όργανα θα πρέπει να προστατεύσουμε το ευρώ αλλά και την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση διότι έτσι έτσι θα πρέπει να αποφύγουμε την δημιουργία εσωτερικών φραγμών και εμποδίων ή στην ε, χρηματοοικονομική αγορά και άρα χρειάζονται χρειάζονται κάποιου είδου εσωτερικέ κινήσει, τόσο να έχουμε τιμολογιακή πολιτική με κάποιε εγγύσει και να έχουμε και την ανακεφαλαιοποίηση. Γιατί αυτό είναι ο χώρο, ο λόγο για τον οποίο θα πρέπει να κάνουμε βήματα προ τα εμπρό. Και έτσι να έχουμε αυτή την κοινή εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο χρειαζόμαστε πιο φιλόδοξη εποπτεία, νομοθεσία των αγορών. Και για αυτό το λόγο θα πρέπει να περισσώσουμε την αξιοπιστία της συντονισμένης μας οικονομικής πολιτικής μέσω της στρατηγικής της Λισαβόνας και την αξιοπιστία του δημοσιονομικού μας πλαισίου στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τώρα, ακούγονται κάποιες φωνές οι οποίες θέτουν το ζήτημα ότι υπό την παρούσα συγκυρία συνεχίδηση η ύφεση στο σύμβολο σταθερότητας θα πρέπει να μπει στο ψυγείο. Δεν είναι όμως αυτό η λύση. Αυτό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Θα πρέπει να τηρηθεί, να συμμορφωθούμε, να εφαρμοστεί. Το 2005 το αναθεωρήσαμε. Εδώ τα συζητήσαμε. Επανειλημμένως όσον αφορά την αναθεώρηση του συμφώνου και τις συνέπειές της. Τώρα έχει περισσότερη ευελιξία των συμφωνών σταθερότητα και είναι στι αντιμετώπιση τη δυσκολία αυτή τη συγκυρία όσον αφορά τα δημοσιονομικά. Όμω, έχοντα αυτή την ευελιξία, το σύμφωνο κέρδισε σε αξιοπιστία. Θα πρέπει να συνεχίσει να απολάβει αυτή τη αξιοπιστία και υπό αυτέ τι συνθήκε και χρειάζεται αυτή η αξιοπιστία, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να εξυπηρετήσουν το δημόσιο χρέο. Με τον καλύτερο τρόπο η αξιοπιστία του συμφώνου επίση χρειάζεται, ούτω ώστε τα spreads να μπορέσουμε να τα συγκρατήσουμε όσον αφορά το δημόσιο χρέο. Επίση, χρειαζόμαστε την αξιοπιστία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια και τι κυβερνήσει να ετοιμαστούν για εξηγήσει δημοσίων να συγκρατήσουν το δημόσιο χρέο αμέσω μετά την έξοδο από το τούνελ τη ύφεση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αλληλέγγυοι προ επόμενε γενναίε. Γιατί έχουμε την πρόκληση του δημογραφικού Επίση, έχουμε την αξιοπιστία του συμφώνου που μας χρειάζεται ούτω ώστε να είμαι θέση θέση να χρησιμοποιήσουν τα δημοσιοοικονομικά, ιδίω τι δημόσιε επενδύσει και δαπάνε στην παιδεία και για μια πιο δυναμική πολιτική απασχόληση, ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε κρίση και να προετοιμαστεί η οικονομία όσο γίνεται συντομότερα για κάποιο είδου ανάκαμψη και εξυγίανση. Ευχαριστώ. Η πρόεδρο, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για όσα μας είπατε. Και με ξεκαθαρίσατε την κατάσταση επί της οποίας, της οποίας βρισκόμαστε, αυτή την ε, πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με αγορά και με το σύμφωνο ε, ανάπτυξη και σταθερότητα. Τώρα, σύμφωνα με την πάγια πρακτική, θα δώσω το λόγο, ούτω ώστε να δούμε τι κάνει το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο τι κάνει για να προχωρήσει προς ένα πλάνο ανάκαμψης. Μπορείτε, μια που είναι εδώ και ο Επιτρόπος φυσικά, να τον ρωτήσετε κάτι και επίσης σύμφωνα με την πάγια πρακτική μας, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Δεν ξέρω αν το κάνετε στα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά εδώ έτσι κάνουμε. Καλά, καλά, ξερούμε στα... Ε, ε, εμείς, κύριος Επίτροπος. Δύο λεπτά. Δύο θα μιλούν τα Εθνικά Κοινοβούλια και ένα Ευρωβουλευτή. Με αυτή τη σειρά θα εναλλάσσονται και τώρα. Για τα Εθνικά Κοινοβούλια, παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σα. Πετε μα πώ ονομάζεστε, ούτω ώστε να ξέρουμε ποιο έχει λάβει το λόγο. Ο πρώτο που έχει εγγραφεί να ομιλήσει είναι ένα συνάδελφο από την Πορτογαλία. Για το Σερά ονομάζεται. Vous avez το λόγο για δύο λεπτά. Και στη συνέχεια θα δώσω σε εσά το. Είστε και εσύ Πορτογάλο. Euh, Ο κύριος ε, του... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ εκπροσωπώ το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο και το μέρος που στηρίζει την ε, Πορτογαλική Δημοκρατία. Και εδώ ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με την παρουσίαση που μόλις έγινε και για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Εδώ, παρόλο που έχουμε πολύ λίγο χρόνο, θα ήθελα να εμπλουτίσω και εγώ την όλη μας συζήτηση με τις ε, δικές μας εμπειρίες. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εξετάζουμε εδώ έχει πολλαπλές διαστάσεις και συνιστώσεις. Βρισκόμαστε στο πέρας μιας οικονομικής κρίσης, χρηματοπιστωτικής, κοινωνικής και πολιτικής. Πρέπει οι Ευρωπαίοι φορείς να σκεφτούν προσεκτικά. Ιδάλλως δεν θα μπορέσουμε να δούμε συνολικά όλα τα συντρέχοντα προβλήματα αυτής της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που παγκοσμίω και στην Ευρώπη έχει ιδιαίτερες συνέπειες. τα προβλήματα που μας απασχολούν σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη συνάντηση, είναι προβλήματα που και η πορτογαλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα, με τρόπο συντονισμένο και με βάση την γενικότερη τοποθέτηση των κρατών μελών ω προς αυτά τα προβλήματα. Όπω ακούστηκε και εδώ, η δράση αυτή πρέπει να είναι συντονισμένη από την πλευρά όλων των κρατών μελών, κατά τρόπο ώστε να υπάρχει αλληλεγγύη και να μην δοθούν, να δοθεί έμφαση στη μια ή την άλλη ταυτότητα κατά τρόπο δυσανάλογο και προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα προστατευτισμού ή ρατσιστικής συμπεριφοράς. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι αυτή η δράση της Ευρώπης πρέπει να εκτελεστεί κατά τρόπο κατά τρόπο ώστε να μην προκληθεί μια πολιτική επίση κρίση. Η πορτογαλική κυβέρνηση, εφόσον βρίσκεται στον ευρωπαϊκό χώρο, έχει κάνει προσπάθεια σε επίπεδο προπολογισμού ώστε να καταπολεμήσει τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης. Έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην απασχόληση και στον δημόσιο τομέα προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία της χώρας. Επίσης, επενδύσεις έχουν γίνει στις πλέον ευάλωτες οικογένειες, κατά τρόπο να αντιμετωπιστούν και τα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν λόγω της κρίσης και κατά τρόπο να εξασφαλιστεί και η σταθερότητα των ε, οικονομικών αγορών. Υπάρχει μια σειρά μέτρων που εκτελεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στην Πορτογαλία, δράσεις οι οποίε ακολουθούν τη γενική γραμμή των ανησυχιών και των υπόλοιπων κρατών μελών. Στόχος είναι να υπάρχει συνοχή μεταξύ κρατών μελών για να μην περάσουμε και σε συνθήκες πολιτικής κρίσης. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο, επειδή είσαστε ο πρώτος που πήρε το λόγο, σα άφησα να μιλήσετε λίγο παραπάνω. Όσο περνάει η ώρα θα είμαι κάπω πιο αυστηρή με το χρόνο. Ο λόγος στον κύριο που ζήτησε λόγο. Από το Ελληνικό Κοινοβούλιο είμαι. Ε, θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Αλμούνια, ε, το οποίο είναι ε, το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θεσμικό επίπεδο για να διευκολύνει τις χώρες οι οποίες δανείζονται με πολύ δυσμενείς όρους σήμερα. Το πρόβλημα είναι γνωστό, αλλά επιτρέψτε μου να θυμίσω το παρελθόν του όταν δημιουργήθηκε το ευρώ γνωρίζαμε ότι υπάρχει το πρόβλημα που οι οικονομολόγοι ονόμαζαν και ονομάζουν ασύμετρα σοκ. και γνωρίζαμε ότι εδώ υπάρχει ένα θεσμικό κενό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω διαβάσει κάποιε δηλώσει του κ. Αλμούνια που υπενήχθηκε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι κοινό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο γύρω από το θέμα αυτό. Δηλαδή εξετάζεται το ενδεχόμενο να εκδοθούν ομόλογα ευρωπαϊκά. Υπάρχουν σκέψεις για άλλους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπιστεί ενδεχομένως και μια κερδοσκοπία η οποία αναπτύσσεται αξιοποιώντας δυσκολίες ορισμένων χωρών να δανειστούν. Αυτό είναι το ερώτημα και θα χαρώ αν μπορούμε να έχουμε κάποια απάντηση. Ευχαριστώ. Και τώρα εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου το λόγο θα λάβει η κυρία Φερέιρα κυρία Ελίζα Φεραίρα, η οποία στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ε, φρόντισε να εγκριθεί η έκτησή τη για το πρόγραμμα ανάκαμψη, όπω ε, τροποποιήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, που θα ε, απασχολήσει ιδιαίτερα βεβαίω στο μέλλον τα κράτη-μέλη. Κύριε Φεραίρα, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε δύο λεπτά θα προσπαθήσω να ανακεφαλαιώσω την τοποθέτηση του Ευρωκοινοβουλίου. Πρώτον, πρέπει να εντοπίσουμε τον κεντρικό μας, τον πρωταρχικό μας στόχο. Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ανάκαμψης είναι η απασχόληση, οι επιχειρήσεις και η τόνωση της πραγματικής οικονομίας. Σε σχέση με αυτούς τους στόχους πρέπει να σταθμίσουμε την επιτυχία ή όχι του προγράμματος της οικονομικής ανάκαμψης πρέπει να πω ότι για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους θα πρέπει να δούμε τριών λογιών θέματα. Πρώτον, τα θέματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, επειδή η πίστοση δεν λειτουργεί όπως περιμέναμε και έπειτα δεν αρκεί. Δεν αρκεί να υπάρχουν πιστώσεις. Χωρίς οικονομική ανάκαμψη η πίστοση είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν είναι επαρκής, είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη. Για να δημιουργηθεί λοιπόν απασχόληση, για να έχουν πρόπτικη για το μέλλον οι επιχειρήσεις, πρέπει να δούμε τι μέσα διαθέτουμε στα χέρια μας. Το πρόγραμμα ανάκαμψης που αποτιμούμε αυτό το διάστημα, όπως υπόθηκε, εκπροσωπεί κατά 15% ευρωπαϊκή, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Το υπόλοιπο είναι οι εθνικές πρωτοβουλίες. Οι χώρες μας έχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων να αντιδράσουν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και πάλι την ατζέντα μας, τις προτεραιότητές μας σε σχέση με την κοινωνική αλληλεγγύη και την εδαφική συνοχή ή με την αρχή της ανταγωνιστικότητας και θα πρέπει να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει με τρόπο σαφή, και αποφασιστικό. Να έχουμε προγράμματα χαρακτήρα οριζόντιου και ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να αξιοποιήσουμε τι διαφορετικέ δυνατότητε των διαφόρων κρατών μελών. Και εδώ ένα μήνυμα που θέλω να απευθύνω στον κύριο Επίτροπο. Λέγεται στην έκθεση αυτή ότι το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει την ετοιμότητά του να περάσει σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο προκειμένου να αναθεωρηθούν οι προτάσεις και οι προτεραιότητες 2007-2013 όπως είχαν προταθεί από την Επιτροπή καθώς και να αναθεωρηθούν τα ανάλογα μέτρα προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος της κρίσης. Αυτό είναι σημαντικό ε, για την Επιτροπή. Δηλαδή μπορεί η Επιτροπή να αξιοποιήσει τα διορθωτικά ταμεία, να ξαναδεί τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν, να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να κινητοποιήσει εγκαίρως τον τομέα της απασχόλησης και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ξεκινώντας προγράμματα οριζόντια, τα οποία να αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που παγκοσμίως αντιμετωπίζουμε σήμερα αλλά και τις ασύμετρες ε, συνέπειες, επιπτώσεις ε, των διαφόρων χωρών, ιδίως όταν ανήκουν στην Νομισματική Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και είναι τα όσα προλάβα να πω σε τόσο λίγο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε άλλη μια σειρά ερωτήσεων. Ο κύριος Μπαλτασάρη πρώτα από την Ιταλία και ύστερα ένα από την Σουηδία και η κυρία Ράιπερ. Ο κύριος Μπάλτας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, καλημέρα σας. Είμαι ο πρόεδρος της, ε, Ευρωπα... της ε, Επιτροπής της Ιταλικής Γερουσίας για θέματα οικονομίας και εμπορίου. Έχω επανεκλεγεί, δηλαδή κατέχω θέση αυτή έξι χρόνια ήδη. Έχω μια ερώτηση λοιπόν δεν πιστεύω και διαφωνώ βαθύτατα ως προς την εκτίμηση ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο μπορεί να αποτελέσει το άθροισμα των επιμέρους εθνικών σχεδίων. Γιατί αυτό το άθροισμα, έστω και συντονισμένο, δεν αποτελεί ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Και κυρίως διότι η κάθε επιμέρους χώρα δρά στο πλαίσιο περιορισμών και ορίων που επιβάλλει η ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Άρα το ερώτημα είναι... Τελούμε γνώση του γεγονότο ότι έχουμε διαπράξει τα τελευταία 4-5 χρόνια δύο τεράστια σφάλματα στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Πρώτο νομισματική πολιτική και ισοτιμία του ευρώ. Και δεύτερο σφάλμα, το ότι δεν αντελήφθημεν ότι ήταν η ώρα να αλλάξει η συνθήκη Μάστεχτ 1 και να περάσουμε στο Μάστεχτ 2 τρέχουσες δαπάνες και επενδύσεις. Το αποτέλεσμα λοιπόν εδώ, αφού ε, φαίνεται ότι μιλάμε μάλλον ακαδημαϊκός πως και όχι πολιτικός, ίσως να σήμαινε και ότι θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη των προβλέψεών μας. Για κάθε ποσοστιαία μονάδα του πληθωρισμού που επιβάλλει μια ελεγχόμενη νομισματική πολιτική έχει και μείωση ως συνέπεια κατά 2% της ανάπτυξης. Και δεν είναι τυχαίο το ότι οι τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, δείχνουν 2% ε, ανάπτυξη λιγότερο και 1% πληθωρισμό αύξηση ε, δηλαδή κάτω από το 2% που είναι ο στόχος. Πάλι η αναλογία είναι 1 προς 2. Αυτές οι εκτιμήσεις, οι προβλέψεις δεν εξαρτώνται από την η ανδήποτε εθνική οικονομική πολιτική, αλλά από την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, η νομισματική καλύτερα πολιτική. Η ανδήποτε εθνική οικονομική πολιτική, τουλάχιστον κατά δύο τρίτα, θα εξαρτάται στο μέλλον από την μεταλλαγή, τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής. Μόνο τότε μπορούμε να μιλούμε για το άθροισμα εθνικών οικονομικών επιλογών. Καλώς, λοιπόν, ευχαριστώ. Η κυρία Μόνικα Γκριν από την Σουηδική Αντιπροσωπεία. Σας ευχαριστώ στα Σουηδικά. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε με την σύγκληση αυτής της συνεδριάσεως. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω και να εκφράσω τις, ε, τα συγχαρητήριά μου για το ε, σχέδιο αυτό Συγκυρία, Ήταν πολύ καλή η λύση που προτάθηκε. Πρέπει τώρα βέβαια να ταθεί σε εφαρμογή χωρίς να εγκαταλείψουμε τη στρατηγική μας. Αντιθέτως πρέπει να εμείνουμε σε αυτά που έχουμε αποφασίσει και να αποφύγουμε την παρέκκληση ή την, ε, ε, τον εκτροχιασμό προς την ε, προστατευτική λύση. Πρέπει να διαφυλάξουμε βέβαια το ελεύθερο εμπόριο, μην προσπαθήσει ο καθένας να προστατεύσει μόνο τις δικές του επιχειρήσεις έναντι των άλλων και να κλείσει τα σύνορά του. Πρέπει να διαφυλάξουμε λοιπόν τις ελεύθερε συναλλαγές αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την αίσθηση της ασφάλεια για τον πολίτης, ώστε αυτός να είναι σε θέση, αισθανόμενος ασφαλής οικονομικά, να προχωρήσει σε επενδύσεις. Αυτό είναι δύσκολο όταν δεν υπάρχει αίσθηση οικονομικής ασφάλειας, όταν κανείς στέκεται ενώπιον οικονομικών ε, ερηπείων, είναι δύσκολο να αναλάβει κανείς οικονομικό κίνδυνο. Πρέπει λοιπόν να ξέρει ο πολίτης ότι ο επενδυτής ότι θα στηριχθεί στην προσπάθεια του αυτή. μέχρι να περάσουν αυτά τα δύσκολα πρώτα χρόνια. Και μετά για, το, για τα μέτρα θα πρέπει να ε, αναλάβουμε, να προβάλλουμε και λύσεις ευφύης, λύσεις σε παραδείγματι αναδιαμόρφωσης ή αναμόρφωσης και των κατοικιών μας ώστε αυτές να γίνουν πιο οικονομικές ε, ενεργειακά, πιο οικονομικές ενεργειακά ώστε να κερδίσουμε σε επίπεδο οικονομικό, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και το περιβάλλον μας, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Λισαβόνα λοιπόν, υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων κατά τρόπο να λειτουργούν αποτελεσματικά και κανόνες μέσω στους οποίους θα προσαρμοστούν όλες οι τράπεζες για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια υγιή οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρέβα Παέβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Βεβαίω και έχουμε πάρα πολύ σημαντικέ ε, προκλήσει. Το αντιμετωπίσουμε λόγω τη ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Ε, είναι κάτι το ο οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και εμείς θα πρέπει ε, να επιδείξουμε ε, θέληση για συνεργασία. Να σας πω ένα παράδειγμα μιας χώρας η οποία απομονωμένη προσπαθεί κάτι να κάνει. Μια χώρα που σχεδόν την γονάτισε. Η χώρα, ε, θα επικαλούμε το πράγμα της Ισλανδίας ταξίδεψα εκεί, μπορώ να σας πω ότι ακόμα ε, δεν ήταν τα χειρότερα, μόλις τώρα άρχισε η κρίση. Εάν όμως η Ισλανδία ήταν μέλος της ΕΕ, αν είχαν λάβει κάποια ταχαία μέτρα, ε, κάποια μέτρα οικονομικής πολιτικής, νομισματικής πολιτικής, δημοσιονομικής πολιτικής, τότε θα είχαν γλιτώσει από πάρα πολλούς μπελάδες. Εγώ ανήκω στους φιλελεύθερους δημοκράτες και ε, θέλω να πω ότι τα κράτη-μέλη για τα σχέδια ανάκαμψης <clears throat> να σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά τους. Είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Επίτροπος. Έτσι θα βοηθήσουν και τις επόμενες γενιές. Δηλαδή, θα πρέπει και αυτόν τον τρόπο να δοθεί μια όθηση στην οικονομία αλλά και στην αγορά εργασία. Βεβαίω και χρειάζονται κάποια άμεσα μέτρα. Όμως χρειάζονται κάποια μέτρα που θα έχουν τελικά μακροοικονομικό αποτέλεσμα και έτσι θα μπορέσει η αγορά να προσαρμοστεί. Ε, οπότε θα πρέπει και αυτόν τον τρόπο να δούμε πώς θα έχουμε κάποιες επενδύσεις σε έργα στην καινοτομία και έτσι να μπορούν οι κυβερνήσεις να ε, κάνουν κάτι. Φυσικά και χρειάζεται κάποιο είδου ρύθμιση, κάποιο είδου νομοθεσία ε, για να βοηθήσουμε επίσης τις ε, επενδύσεις. Να μας πούνε γιατί πιστεύουν οι συναδέλφοι τα Εθνικά Κοινοβούλια και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να δημορφώσουμε μια κοινή θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων πέρασε ένα ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο προτείνουμε την μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Ακόμα, επομένως, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Επίσης υπάρχουν για τον ΦΠΑ δύο θεωρίες, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι η μία αντιβαίνει στην άλλη. Τώρα λέει διαφοροποίηση και τώρα λέει μείωση των συντελεστών. Οπότε οι παράγοντες που πρέπει να υπόψη είναι η ανταγωνιστικότητα, η διαφάνεια, αλλά και η καλύτερη ευκολότερη διαχείριση του φορολογικού συστήματος. Εσείς κύριε Επίτροπε τώρα πέστε μας, τι διδαχθήκατε από την χρηματοοικονομική κρίση. Και πάλι ένας ε, συνάδελφος από την Πορτογαλία, κύριος Νέτου, μετά ένας συνάδελφος από τις κάτω και μετά ο κύριος Χινάς. Ζόρζο Νέτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι Πρόεδρος της Δημοσιονομικής και Οικονομικής Επιτροπής του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου. Γνωρίζω πολύ καλά τον κύριο Αλμούνια από όταν ήταν, από όταν ήταν πρόεδρος της ε, ομόλογης Επιτροπής του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Είναι χαρά μου λοιπόν που τον ξανασυναντώ σήμερα εδώ. Τώρα το ερώτημα που ήθελα να του απευθύνω είναι ένα ερώτημα πραγματιστικό και περί μεθοδολογίας για το πρόγραμμα ανάκαμψης, οικονομικής ανά, ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά την μεθοδολογία μας, διότι στο παρελθόν έγιναν αρκετές απόπειρες να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα που δεν απέβησαν όμως ε, επιτυχής. Θυμίζω το πρόγραμμα του κ. Πόλσεν στις Ηνωμένε Πολιτείες που αρχικά σκοπό είχε να καταπολεμήσει τα αρχικά προβλήματα της κρίσης, ενώ στη συνέχεια πέρασε στην αντιμετώπιση των κεφαλαιοχικών προβλημάτων των τραπεζών. Σήμερα προτείνεται ένα νέο πρόγραμμα, γιατί το πρόγραμμα Πόλσεν έδειξε ότι ήταν αναποτελεσματικό και λοιπέ προκειμένου να αντιμετωπίσει τι επιπτώσεις της χρηματοποστατικής κρίσης. Και στη Μεγάλη Βρετανία είδαμε ο Πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν υπέβαλε ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρήθηκε αρκετά καινοτόμο για επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για εγγύσει προς τι τράπεζε ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Όμως αναγνωρίζεται σήμερα ότι και στη Μεγάλη Βρετανία χρειάζεται άλλο πρόγραμμα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Γι' αυτό διαρωτώ με κατά πόσον το πρόγραμμα ανάπτυξη, ανάκαμψης, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το πλέον εύστοχο για να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση. Και διαρωτώ με, γιατί νομίζω πρέπει να σκεφτούμε ακόμη πιο προσεκτικά για την κατάσταση, για το πώς έχει και τις διαστάσεις της κρίσης πριν υποβάλουμε ένα πραγματικό πρόγραμμα ανάκαμψης. Να θα θυμίσω ότι κατεξοχήν υπάρχουν παραδείγματα, καταστάσεις παραδειγματικές όπως αυτές της Σουηδίας, η κρίση της Σουηδίας, που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη σε σχέση με το παρελθόν. Η Σουηδία σε πρώτη φάση προέβλεψε ένα πρόγραμμα μελετώντας προσεκτικά την τραπεζική κρίση Πρώτα έγινε σοβαρή εξέταση του φαινομένου και μετά υπευλήθη πρόγραμμα. Πρόγραμμα επιτυχημένο για να αντιμετωπιστεί η κρίση στη Σουηδία. Η κρίση του χρηματοπιστωτικού και οικονομικού συστήματος. Έτσι πρέπει να δούμε και το παράδειγμα της Ιαπωνίας όπου υπήρξε τραπεζική και χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα με τον καταλληλότερο τρόπο. 20 χρόνια αργότερα Υπάρχει ακόμη σοβαρό πρόβλημα που εμένει, διότι δεν έγινε προληπτικά και προηγουμένως ενδελεχής σοβαρή προσεκτική ανάλυση της πραγματικής κατάστασης των τραπεζών στην Ιαπωνία και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Γι' αυτό λοιπόν αναρωτιέμαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς έχουμε κάνει το έργο μας προηγουμένως εκ των προτέρων ξέρουμε ποιε είναι οι διαστάσει τη χρηματοπιστωτική και τραπεζική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχουμε μελετήσει τι διαστάσει πριν υποβάλουμε το πρόγραμμα ανάκαμψη. Διότι αν δεν ξέρουμε τη διάσταση και το βάθο τη κρίση, το πρόγραμμα αυτό νομίζω είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Και δυστυχώ δεν θα έχει την επιτυχία που προφανώ εμεί ελπίζουμε και αναμένουμε διακαώ στι χώρε μα. Ευχαριστώ. Δεν θα τολμήσω να είμαι τόσο αυστηρή και εγώ με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά θα σας παρακαλέσω ξανά να σεβαστείτε το χρόνο ομιλία σας. Πιο αυστηρή θα με τους συναδέλφους από το Ευρωκοινοβούλιο μόνον. Να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο από την Ιρλανδία. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο Ιρλανδούς συναδέλφους θα πάρει το λόγο, παρακαλώ να συστηθείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Φαντάζομαι και εμείς έχουμε τα δικά μας προβλήματα, τα διόρυθμα, μια που είναι ανοιχτή η, η οικονομία μας κατέρευσε δε και η φούσκα όσον αφορά τα ακίνητα. Εθνικοποίησαμε τράπεζες, αν επανακεφαλαιοποίηση γίνεται στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα. Ε, θα γίνει συγκράτηση μισθών και τιμών και δαπανών όσον αφορά τη δημοσιοτομία. Φυσικά και αντιλούμε μαθήματα από τους ε, άλλους στην Ευρώπη για το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Πάντως, όντως θα πρέπει να κάνουμε ε, επενδύσεις στην ενέργεια και στην καινοτομία που άλλωστε πάντοτε μας απασχολούσε ο κλάδος Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην Ευρώπη και γι' αυτό ήρθαμε και σήμερα να μάθουμε το αύριο. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε πιο αποτελεσματική νομοθεσία στο χρηματοοικονομικό τομέα χωρίς βέβαια να τον φημώσουμε αυτόν τον τομέα γιατί και αυτός ο τομέας και αυτός ο κλάδος θα βοηθήσει τόσο ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από το αδίεξοδο. Ευχαριστούμε πολύ, Λέω Πρόεδρος. Και τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριο Χίνα, για λογισμό των χριστιανοδημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την αντίδραση από την κρίση ασχολούμαστε με την αντίδραση για έξοδο από την κρίση, αλλά νομίζω, Επίτροπε, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πρόληψη. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξανασυμβεί ποτέ αυτό που οι πολίτες υποφέρουν σήμερα στην καθημερινότητά τους το πρόβλημα η ασυμμετρία είναι γνωστή ότι σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη οικονομία τα κεφάλαια οι ροές είναι υπερεθνικές και η λογοδοσία και ο δημοκρατικός έλεγχος όπου αυτός υπάρχει είναι εθνικός. Αυτή είναι η μεγάλη ασυμμετρία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη την πάθαμε μια φορά. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην την ξαναπάθουμε εσείς ως εκπρόσωπος της ευρωζώνης και της ε, ε, ορθοδοξίας στην πολιτική της ονέ κάνετε άριστα τη δουλειά σας αλλά ξέρετε πολύ καλά όπως ξέρω κι εγώ ότι υπήρχαν άλλοι παίκτες στο κανονιστικό παιχνίδι που απέτυχαν να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι αυτοί που ήλπιζαν ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα αυτορυθμιστεί είναι αυτοί οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών οι οποίοι δεν είδαν το παγόβουνο να έρχεται πάνω στον τιτανικό αλλά μετά είδαν πολύ εύκολα τις χώρες που είχαν προβλήματα δανεισμού. πρέπει λοιπόν επίτροπε εκτός από την νομισματική ορθοδοξία της ευρωζώνης την οποία εκφράζεται και την οποία θα συνδράμουμε όπως μπορούμε και από το ευρωπαϊκό και από τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να μας διαβεβαιώσετε ότι το κανονιστικό πλαίσιο που θα αποτρέπει τέτοιες καταστροφές στο μέλλον θα υπάρξει και θα είναι επαρκές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει τώρα η δανική αντιπροσωπεία. Δεν ξέρω δηλαδή ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος ο οποίος θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι ο αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής Οικονομικών και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Έχουμε τώρα μία πολύ ισχυρή κατάσταση ε, και γι' αυτό έχουμε οπλιστεί και σωστά και είμαστε σε καλύτερη θέση από ό,τι άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή μπορούμε ε, να επιβιώσουμε πολύ καλύτερα από την λέλαπα ε, την οποία αντιμετωπίζουμε και έχει αποδειχθεί ότι τα ε, οι πιστώσεις ε, στο σύστημα έχουν παγώσει και εμείς στη χώρα μας έχουμε επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα πιστώσεων για να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση και διαπιστώνουμε ότι λειτουργεί σωστά. Στην ε, Δανία έχουμε επίσης επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα αναπτύξεως αλλά πρέπει συγχρόνως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί στη Δανία πρέπει να προσπαθήσουμε να να μην κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις. Ε, θα πρέπει να επιλέξουμε το σωστό σημείο για να ε, ε, επέμβουμε διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να είναι αποτελεσματικό και οποιοδήποτε πρόγραμμα εφαρμόσουμε για την οικονομική ανάκαμψη. Θα θέλαμε λοιπόν να πούμε ότι μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να προσπαθήσουμε να κινηθούμε από κοινού και να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση και να προσπαθήσουμε ε, να ε, αντεπεξέλθουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Σαλμούνια είναι πολύ βασικό. Δεν θα πρέπει να υπερισχύσει ο προστατευσισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η σύγχρονη Ευρώπη την οποία προσπαθούμε να να οικοδομήσουμε εδώ και χρόνια να ε, μην ξαναγυρίσει στην εποχή των ατομικών πολέμων όπου έπρεπε ο καθένας να φροντίζει για τα του οίκου του. Ε, πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να διατηρηθεί σε σωστή κατάσταση και όσο αναφορά το δανέζικο μοντέλο της, ε, του συνδυασμού ευελιξίας με ασφάλεια, flex security, θα έπρεπε να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, διότι δίνει μεγαλύτερη ε, ασφάλεια στην αγορά εργασία και μπορεί να επηρεάσει θετικά. Ακριβώς ε, αυτή η ε, άποψη θα πρέπει να υπερισχύσει και σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Κόνραντ από την Αυστρία και είμαι ο, πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Αυστρίας. Θα έπρεπε εδώ να μπορέσουμε ε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση πιο σφαιρικά και δεν μπόρεσαν οι υπεύθυνοι να ε, ασχοληθούν με την κατάσταση κατά αυτόν τον τρόπο γι' αυτό και είχαμε τόσες πολλές ζημιές στις τράπεζες στο μέλλον και εδώ σας είμαι πολύ ευγνώμων κύριε Πρόεδρε διότι νομίζω ότι εσείς ε, πρεσβεύετε ε, την λήψη και πολιτικών μέτρων μέχρι στιγμής έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά μέτρα για να μπορέσει να αντεπεξέλθει της κρίσης και υπάρχει ένα πακέτο πακέτο στη χώρα μας 3,5 δισεκατομμυρίων μαζί με άλλα προγράμματα και με την τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε καλύψει το 2,5% του ΑΕΠ για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε της κρίσεως. Θα ήθελα να πω και κάτι ολοκληρώνοντας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ κατά τη διάρκεια της κρίσεως θα πληγεί περισσότερα και δεν θα πρέπει να έχουμε προβλήματα με τις θέσεις εργασίας στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γι' αυτό και ζητώ να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να μπορέσουν αυτές οι μικρές ε, επιχειρήσεις ε, να διατηρηθούν και να ευημερήσουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα, Θα δώσω τώρα το λόγο στους Έλληνες συναδέλφους για τον επόμενο γύρω. Την κυρία Βαντενμπρουκ. Θα ζητήσω βέβαια από τον Επίτροπο να απαντήσει σε το τον πρώτο κύκλο. Κυρία Βαντενμπρουκ, λοιπόν. Πρώτα. Βαντενμπρουκ. Το θέμα στο που θέλω να αναφερθώ το έχετε και εσείς πιστεύω θίξει στην ομιλία σας. Το ακούσαμε και στην έκθεση της κυρίας Φερέιρα. Γιατί δυστυχώς δεν υιοθετήθηκε με την ίδια αυτή διατύπωση σήμερα κατά την ψηφοφορία. Πρόκειται για το θέμα των αξιογράφων στις ε, διάφορες χώρες μέλη, κυρίως των ομολόγων που έχουν μεγάλη ανάπτυξη στα κράτη-μέλη με μια προσπάθεια μάλιστα να αναπτυχθούν και ε, ομόλογα κοινά μεταξύ είτε διαφορών περισσότερων κρατών είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θέλουμε να δούμε εάν θα έχουν αυτά όχι διαφορετικό τόσο αποτελέσμα όσο προσθετικό αποτέλεσμα, εάν μπορούν κάπως να βοηθήσουν στην προσέλκυση περισσότερων κεφαλαίων και δι έξω από την Ευρώπη, προχωμένων από χώρες εκτός της Ευρώπης. Διότι βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν έλλειμμα του 10% αλλά και μεγαλύτερο ακόμη μερικές φορές, είναι όμως σε θέση χάρη στα ε, ομοσπονδιακά του ομόλογα να προσελκύσουν από τι διεθνεί αγορές πολύ περισσότερα κεφάλαια από ό,τι μπόρεσε να ε, εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν αρκετοί δισταγμοί σε επίπεδο συμβουλίου ω προ την εξέταση ακόμη και αυτής της προοπτικής. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν και από τους άλλους συναδέλφους και ιδίως από τα εθνικά κοινοβούλια τι βλέπουν εκείνοι και βέβαια και την Επιτροπή να μας πει αν έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για τέτοιου είδους ομόλογα ή αν έχει πληροφορίες γενικότερες, αριθμητικά στοιχεία, στατιστικές, εκτιμήσεις ενδεχομένως πώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με το μέσο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Όπως βλέπετε, οι εθνικοί βουλευτές και οι ευρωβουλευτές σε πολλά σημεία συγκλίνουν ως προς τις θέσεις τους. Ας ακούσουμε λοιπόν τις απαντήσεις και μετά τον επόμενο γύρο ερωτήσεων και πρώτος θα είναι ο πρόεδρος κύριος Αγοραστός, μετά ο κύριος Λιμίνη από την Ιταλία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. συμφωνώ με πολλές από τις ε, παρατηρήσεις που ακούστηκαν, από τις ερωτήσεις, τις παρεμβάσεις σας. Συμφωνώ πλήρως δε με εκείνους οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη για ενίσχυση του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συντονισμός σημαίνει περισσότερη αποτελεσματικότητα ως προς τα αποτελέσματα των πολιτικών, των μέτρων δηλαδή που υιοθετούμε. Συντονισμός σημαίνει ταυτόχρονα όμως και τον εκτονώνου κάνευ όρο για την πιο ισοδίκαιη κατανομή των προσπαθειών. Συμφωνώ πλήρως με όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι η Ευρώπη σε αυτούς τους δεινούς καιρούς χρειάζεται την αλληλεγγύη των μελών της. στην Ευρώπη έχουμε πολιτικές συνοχές, συνοχής που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους. Προσπαθούν να αντισταθμίσουν κάποιες από τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσεως. Προετοιμάζουμε και ε, προτάσεις που αυτή τη στιγμή συζητεί τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτάσεις οι οποίες θα εξασφάλιζαν πιο ευέλικτη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής για να επαναπροσδιοριστούν προτεραιότητες, εάν είναι αυτό απαραίτητο, στα προγράμματα και τις επενδύσεις που χρηματοδοτούν αυτά τα ταμεία. Και κάποια κρατημέλη εργάζονται σκλήρα στον στόχο του επαναπροσδιορισμού αυτών των προτεραιοτήτων. Εχθέ είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με έναν Υπουργό των Οικονομικών, ο οποίος με ενημέρωσε για το πώς η χώρα του το έργο αυτό το έχει ξεκινήσει ήδη, ένα έργο πολύ χρήσιμο, απαραίτητο σε αυτή την εποχή και όντως διαπιστώνουμε ότι η ελεγγύη θα πρέπει να ξεπεράσει την απλή ε, αποτελεσματικότητα των μέσων συνοχής. Γιατί αλληλεγγύη σημαίνει ταυτόχρονα και αποτροπή του προστατευτισμού στις διεθνείς αγορές, αλληλεγγύη σημαίνει ταυτόχρονα και κοινό όραμα και όχι μόνο το συνοθήλευμα των επιμέρους οραμάτων. Κάποιοι αναφέρθηκαν στον ΦΠΑ και τα ποσοστά του ΦΠΑ. Ε, ακούστηκαν προτάσεις για μείωση ε, για, ε, για ορισμένα προϊόντα προτεραιότητας των ποστών του ΦΠΑ, επί παραδείγματι για υπηρεσίες έντασης εργασίας ή για δραστηριότητες οικολογικού αποτελέσματος, πράσινες λεγόμενες δραστηριότητες. Και σας διαβεβαιώ ότι τις συζητήσεις αυτές τις διεξάγει σε επίπεδο ΕΚΟΦΗΝ το Συμβούλιο με ιδιαίτερα επώδυνες συνθήκες διότι χρειάζεται η ομοφωνία των 27 δηλαδή υπουργών των οικονομικών προκειμένου να τροποποιηθεί η ελάχιστη τελεία από την οδηγία αυτή για την, για το, για την φορολογία στο ΦΠΑ και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι το καλύτερο για τη σημερινή εποχή. Χρειαζόμαστε κοινέ δράσει και κοινέ αποφάσει για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Και ίσω μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα και τα φορολογικά μέσα στην προσπάθεια αυτή. Συμφωνώ επίση με τι παρατηρήσει που αφορούν τι προτεραιότητε για τι επενδύσει, με τα διαρθρωτικά ταμεία, με του εθνικού προπολογισμού, αλλά ταυτόχρονα και με του πόρου που εξασφαλίζει η δανειοδοτική δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και θα δείτε τον κύριο Μάιστατ, θα ακούσετε μάλλον τον κύριο Μάιστατ σε λίγα λεπτά, ε, ορίζουμε λοιπόν νέες προτεραιότητες και στις επενδύσεις σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας για τις κλιματικές αλλαγές. Εδώ είναι η παριθμόν ένα προτεραιότητα πάνω απ' όλα και έχουμε ταυτόχρονα να κάνουμε και με ένα πολύ ισχυρό μέσο που μπορεί να υποστηρίξει τις οικονομίες μας την ανάκαμψη, την οικονομική πάνω απ' όλα ανάκαμψη το ταχύτερο δυνατό. Δεύτερη παρατήρηση. η χρήση στην προσπάθεια για την επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων των ε, κυβερνήσεων, των κρατών, του δημόσιου τομέα δηλαδή των χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι αγορές πιέζουν περισσότερο τις κυβερνήσεις. Τα ομόλογα, τα κρατικά ομόλογα, τα spread έχουν ανοίξει. Σε πολλούς μάλιστα τομείς των χρηματοπιστωτικών αγορών βλέπουμε ότι τα spread έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από ότι τα κρατικά ομόλογα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξοδε από τη ζώνη του ευρώ. Είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκάστηκαν να καταβάλουν υψηλότερο spread από το ύψιστο που γνώριζε η ζώνη του ευρώ. Αυτό που έχει τώρα η Ελλάδα με την Ιρλανδία μαζί. Αυτή η πίεση λοιπόν των αγορών αποτελεί πιστεύω και απόδειξη ή ένδειξη της ανησυχίας που αισθάνονται οι αγορές και που έχω επισημάνει τις τελευταίες εβδομάδες αρκετές φορές ότι είναι μηδέν η πιθανότητα να διαραγεί η ζώνη του ευρώ. Όχι 0,1, είναι 0, απόλυτο 0. Δεν υπάρχει τόσο να διαραγεί η ζώνη του ευρώ. Δεν διανοούμε κυβέρνηση να αποφασίσει κάτι τέτοιο. Είναι αδύνατο για λόγους λογικούς, όχι γιατί, δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν νομικοί περιορισμοί. Για λόγους λογικής ορθολογισμού δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο των αντίον κάθε μέρα βλέπω να επεκτείνεται και ο κατάλογος των υποψηφίων για την ένταξη των ζώνη, ζώνη του ευρώ η Ισλανδία που αναφέρατε κάποιοι η Ισλανδία ζητά να μπει στη ζώνη του ευρώ πριν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το πάει ανάποδα. Προσπαθεί να μπει στη ζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με κύριο στόχο να μπει στο ευρώ το ταχύτερο δυνατόν. Και δεν είναι και η μόνη. Πολλέ άλλε χώρε και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνω δε ότι κάποιε από αυτέ ήταν πολύ επιφυλακτικέ μέχρι και πολύ πρόσφατα ω προ τα πλεονεκτήματα τη ζώνη του ευρώ. Και τώρα δια, διακαώ επιθυμούν την προσχώρηση. Κάθε χώρα έχει πιστοτικό κίνδυνο, τον οποίο καταμετράμε χάρη στο spread. Το spread σήμερα υπερεκτιμά πιστεύω τους πιστοτικούς κινδύνους, αλλά ενδέχεται όταν οι αγορές συναλλάσσονται σε κρατικά ομόλογα ή σε ή όταν γίνεται αυτή η κυκλοφορία των κρατικών ομολόγων να προσαρμοστεί στον ε, κίνδυνο αυτόν το spread. Πάνω από όλα αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης, της κάθε χώρας που πλήττεται από το μεγάλο αυτό spread. Γιατί δηλαδή σε ορισμένες χώρες είναι πιο υψηλό το spread από ό,τι σε άλλες. Την ερώτηση λοιπόν πρώτα απ' όλα θα την δώσουν οι αρχές της χώρας, όχι οι ευρωπαϊκές αρχές. οι ευρωπαϊκές αρχές συμβάλλουν στην ομαλή εκτίμηση του κινδύνου. Και αυτό το κάνουμε λογικά και με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και με τις και εκτιμώντας τις δράσεις των αρχών που ε, εργάζονται ε, για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και των, των πολιτικών της ζώνη του ευρώ. Πάνω απ' όλα όμως, όπως είπα, η ευθύνη είναι των αρχών των κρατών μελών. Οι δε πολίτες των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι για να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κερδίσει πλεονεκτήματα, όντας δηλαδή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κερδίσει πολλά πλεονεκτήματα, κερδίσει πλεονεκτήματα η χώρα τους, αλλά φέρουν και μεγάλε ευθύνε. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. σε ποιο βαθμό θα ήταν καλή ιδέα η έκδοση ευρωπαϊκού ομολόγου, ομολόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα. Πλην όμω, δυστυχώς, μη βιώσιμη τώρα λόγω των συνθήκων των αγορών. Τώρα δεν θα είχαμε κράτη-μέλη ή κάποια κράτη-μέλη κρίσιμη σημασία για την έγκριση μιας τέτοια άποψη ε, ενός τέτοιου μέτρου. Δεν θα μα υποστήριζαν, δηλαδή κάποια κρίσιμα κράτη-μέλη προς το παρόν. Για λόγους οικονομικών συνθήκων, για λόγους συνθήκων στην αγορά. Πλην όμως, εμείς θεωρούμε ότι είναι καλή ιδέα συνεργίζουμε την επεξεργασία τη. Υπάρχουν κράτη-μέλη που συμμετέχουν και συνεργάζονται μαζί μα, θέλουν να συνεργαστούν μαζί μα στην προώθηση ιδέα αυτή, αλλά δυστυχώ δεν είναι κατάλληλη η στιγμή για την υιοθέτηση ενό τέτοιου μέτρου. Είναι όμω κατάλληλη στιγμή να υιοθετηθούν εναλλακτικέ λύσει ίσως όχι τόσο καλές, αλλά πάντως βιώσιμες μακροπρόθεσμες. Μακροπρόθεσμα τις έχουμε συζητήσει. Επί παραδείγματι προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να συντονίσουμε καλύτερα μια τέτοια έκδοση δεδομένων των κρίσεων της αγοράς, δεδομένων των νέων εκδόσεων κρατικών ομολόγων που έχουν προεξαγγελθεί για το 2009. Αλλαγές στην ευρωπαϊκή πολιτική ή σε ποιο βαθμό η ευρωπαϊκή πολιτική έχει ευθύνη, είναι συνυπεύθυνη για τόσα συνέβησαν. Μα κοιτάξτε όμως, τόσα συνέβησαν δεν έχουν συμβεί μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι ΗΠΑ και στην ε, Ιαπωνία και την Νότια Κορέα. Σε κάθε χώρα, σε κάθε οικονομία του κόσμου εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα. Μην ρίχνετε το φταίξιμο στην Ευρώπη για την εμφάνιση μιας της παγκόσμια κρίση. Εάν πρέπει να βρούμε κάποιον υπέτειο, μακροοικονομικά υπέτειοι είναι αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν της σε παγκόσμιο επίπεδο ανισορροπίες. Ευχαριστώ να γίνω και πιο συγκεκριμένο εάν το επιθυμείτε. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι προκάλεσαν τις ανισορροπίες παγκόσμιες στις οικονομίες μας. Αυτό είναι, είναι γνωστοί ποιοι είναι αυτοί. Και από μικροοικονομική σκοπιά η πέτη είναι εκείνοι οι οποίοι υπεστήριξαν την μη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, τη μη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, τη μη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και των ε, rating agencies. Εκείνοι οι οποίοι χάρη σε αυτή την κερδοσκοπική ε, στάση κέρδισαν, κεροσκόπησαν, κέρδοσκόπησαν πάνω σε αυτό το σύστημα, σε αυτήν την ανισορροπία. Μην ρίχνετε ως το φταίξιμο σε εκείνους που υποστήριζαν τη ρύθμιση, την νομοθεσία, τον έλεγχο. Και επίσης ένα άλλο σημείο. αναλογισμός και αντίδραση ως προς την χρηματοπιστωτική κρίση, την κρίση χρηματοπιστωτική. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, το μελετούμε διαρκώς, ε, θα καταθέσουμε προτάσεις, επεξεργαζόμαστε εν ώψη και του G20 και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μαζί με την ομάδα Ντελαρόση κάνουμε προτάσεις, ε, θα, θα κάνουμε καλύτερα προτάσεις μετά την υποβολή τη της εκθέσεως της ομάδας Πλην όμως... Η πολιτική απόφαση, η επιλογή του αν θα πρέπει να δράσουμε, να υιοθετήσουμε λύσεις πριν από την εξασφάλιση μιας σφαιρικής εκτίμησης της κρίσης, από μένα λαμβάνει καταφατική απάντηση. Εγώ λέω δεν έχουμε περιθώριο να περιμένουμε περισσότερο. Και όπως είπε και ο νέος πρόεδρος των Οικονομικών της ΗΠΑ εχθές, όταν παρουσίασε στη Washington τις νέες προτάσεις, το νέο πακέτο προτάσεων για την στήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα, Είπε λοιπόν ο Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ ότι ίσω να μην είναι το τελευταίο πακέτο, ίσω κάποια από τα μέτρα που περιλαμβάνει να μην λειτουργήσουν αποτελεσματικά, ίσω να χρειαστεί να προσαρμοστούν τα μέτρα αυτά στο μέλλον. Πλην όμω είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να λάβουμε τα μέτρα, διότι αν δεν το πράξουμε, ο κίνδυνο τη κατάρρευση συνολικά του οικονομικού τομέα που αποφύγαμε τον Οκτώβριο μπορεί πάλι να επανεμφανιστεί. Και δεν έχουμε περιθώριο για τέτοιου είδους επανεμφάνιση, για τέτοιο κίνδυνο. Για δε τον πολίτη, για δε την ε, σκοπιά της πραγματικής οικονομίας, αντιλαμβάνομαι, εγώ είμαι και πολίτης, δεν είμαι μια χρηματοπιστωτική αγορά, πολίτης είμαι πάνω απ' όλα, αντιλαμβάνομαι πλήρως το επιχείρημα παρακαλώ μη δίνετε τα λεφτά σε αυτούς που προκαλέσανε την κρίση, δώστε μου εμένα τα λεφτά απευθεία στον πολίτη. Αλλά το να χορηγήσω κονδύλια, το να δώσω πόρους στον πολίτη, την επιχείρηση, την εταιρεία, προϋποθέτει ότι θα έχω και τη χρηματοπιστωτική αγορά. Τη χρειάζομαι τη χρηματοπιστωτική αγορά. Αυτή θα διαθέσει, θα κατανείμει, θα δανείσει το χρήμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια στέρη, μια υγεία, μια φερέγγια χρηματοπιστωτική αγορά, αλλά χρειαζόμαστε και χρηματοπιστωτικέ δραστηριότητε. Και έτσι πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να παρακολουθήσουμε, όπω άλλωστε και τώρα, τι δραστηριότητε του χρηματοπιστωτικού τομέα, τι υπηρεσίε εκείνε οι οποίε δεν λειτουργούν όπω πρέπει. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων μέχρι να έρθει μαζί μας ο επόμενος καλεσμένος μας. Πάντως να αντιδράσω εγώ ίδια στην τελευταία σας παρατήρηση. Να πω ότι εάν η τραπεζική αγορά και αυτή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν λειτουργεί, αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει πρόβλημα και με την οικονομία. Τώρα, αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, είναι κάτι άλλο. Πρέπει να, λειτουργούμε και προ τι δύο κατευθύνσει και να τι εξετάζουμε και τι δύο. Διότι η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό κλάδο πρέπει να ανακτηθεί. Αλλά η σταδιακή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σαφώ δεν πρέπει να επικεντρωθεί σε ένα και μόνο μέτωπο. Δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση στην κοινή γνώμη των χωρών μα ότι ανησυχούμε μόνο για τον τραπεζικό κλάδο. Και μια δεύτερη παρατήρηση. Αρχίζουν πλέον να, να λύνονται οι γλώσσε. Και πλέον μιλάμε ανοιχτά. Βλέπουμε ότι η στήριξη προς τις τράπεζες ε, προτάθηκε αρχικά και αποφασίστηκε και προωθήθηκε Πρώτον, σε κλίμα πανικού, βλέποντα ότι υπάρχει κρίση με τη φερεγγιότητα του συστήματο, αλλά κάποιε φορέ και χωρί πολλέ-πολλέ διαπραγματεύσει δεν ήταν ο σκοπός ε, να περάσει κανείς σε πλήρεις ε, νομοθετικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Όμως κάποιοι από εμά πλέον πιστεύουν ότι έπρεπε να έχουν τεθεί, κάποιοι, να έχουν τεθεί κάποιες προϋποθέσεις τη στιγμή που χορηγεί το, η βοήθεια προς τις τράπεζες. Και τώρα ξεκινάει και η συζήτηση για κάτι που θα μπορούσε να ονομαστεί ως τρίτο επίπεδο. Μετά τις τραπεζικές εγγυήσεις, την επανακεφαλαιοποίηση, μιλάμε πλέον για τοξικά προϊόντα, μιλήσαμε για τοξικά προϊόντα και τώρα μιλάμε και για ακάθαρτα προϊόντα. Άρα αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει τώρα είναι η υλοποίηση του τρίτου αυτού του τρίτου όπως ονομάζεται όροφος. Ε, μπορώ να τη δράσω με το πρόνομο του Επιτρόπου στα λεγόμενά σας. Ναι, υπάρχει αυτή η διάδραση που αναφέρατε μεταξύ από τη μια της στήριξης, δηλαδή της μείωσης του επίπεδου χρέωσης, που είχε ξεπεράσει το επίπεδο του λογικού και της απονομής κονδυλίων για τη δημιουργία νέων πιστώσεων, για την χρηματοδότηση νέων δραστηριοτήτων που θα δώσουν νέα όθηση στην, ε, στην οικονομία. Τη μη χρηματοπιστωτική οικονομία που θα της επιτρέψουν να ανακτήσει το δυναμικό της χαρακτήρα. Ε, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει διάδραση και αλληλεπίδραση. Όμως, εάν πρέπει να ξεκινήσουμε από το ένα από τα δύο άκρα της πορείας αυτής, θα πρέπει νομίζω να ξεκινήσουμε από τη μη χρηματοπιστωτική οικονομία με προγράμματα ανάκαμψης και νομισματικές πολιτικές αρκετά πιο εκτατικές σε σχέση τουλάχιστον με το παρελθόν, αλλά βλέπουμε ότι αυτό που έγινε από την πλευρά της αίτηση, της ζήτησης δεν θα λειτουργήσει, δεν θα πιάσει εάν συνεχίσουμε να μην αναλαμβάνουμε μέτρα και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορεί. Υπάρχει λοιπόν δίλημα. Τίθεται δίλημα. Δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς. Για τα πληγέντα στοιχεία, αυτά που έχασαν την αξία τους, ε, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τα τοξικά ενεργητικά όπως ονομάζονται, αλλά και με τα μη τοξικά που μπορεί όμως να γίνουν τοξικά στο μέλλον, εάν δεν βρεθεί λύση εγκαίρως. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διαπραγματεύσεις, ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι πρέπει να οριστούν όροι, όροι και συνθήκες για να κατανεμηθεί σωστά ο φόρτος ή κίνδυνοι όταν μιλάμε για το χρήμα του φορολογουμένου ή όταν χρησιμοποιούμε τη συμβολή των ε, φορολογουμένων για να αναχαιτήσουμε προβλεπόμενους κινδύνους. Αυτές είναι συνθήκες, είναι όροι που πρέπει να τεθούν επιτάπητος. Κάποιες χώρες το έκαναν ήδη αυτό, προβλέπεται στα προγράμματά τους, άλλοι σε λιγότερο βαθμό. Όμως, κατά την άποψη της Επιτροπής, είναι μια σαφής προϋπόθεση για να έχουμε οικονομική επιτυχία όχι μόνο για την πολιτική μας επιτυχία, για την ίδια την οικονομική επιτυχία αυτή καθ' αυτή. Γιατί αλλιώ ε, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς θα τους δώσουμε την εντύπωση ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και ότι το κράτος και οι φορολογόμενοι μια ζωή θα τους διασώζουν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Αγοραστό και έπειτα από την Ιταλία ο κύριος Τζορτζέτη και μετά από το Ευρωκοινοβούλιο κυρία Μπατζελή. Ο κύριος Αγοραστό. Πρέπει να επισημάνουμε ότι κανένα πρόγραμμα, κανένα μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Συνεπώ χρειάζονται μέτρα υπέρ των πολιτών και χρειαζόμαστε τη συμμαχία των πολιτών για να ξεπεραστεί η κρίση μέσω των δημοσιονομικών μέτρων αλλά και των νομισματικών πολιτικών. Ακόμη πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και η παγκοσμιοποίηση αποτελεί φαινόμενο επιτάχυνση της οικονομίας σε όλα τα επίπεδα. Η επιτάχυνση αυτή διευρύνει τις συνέπειες των κρίσεων εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι εκτικοί μηχανισμοί. Και ναι βέβαια οι αγορές είναι ένα εργαλείο δημιουργίας πλούτου, αλλά όταν δεν υπάρχει εποπτικό μάτι βγαίνουν εκτός ελέγχου με τις συνέπειες τις οποίες βλέπουμε σήμερα. Είχαμε δει με μικρότερη ένταση πριν τέσσερα χρόνια τη φούσκα ε, του ίντερνετ και πριν από 8 χρόνια τη φούσκα ε, των κατασκευών. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι αποτέλεσμα της ασύμετρης πληροφόρησης. Άρα πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση των επενδυτών και των εμπλεκομένων μελών που οδηγεί σε επαχθείς επιλογές για επενδυτές στο πλαίσιο του κινδύνου χαλάρωσης της διοντολογικής ηθικής μέρημνας ο οποίος έφτασε στα επίπεδα πλεονεξίας. Συνεπώς δεν υπήρξε επαρκή ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Επίσης υπόθηκε για τον ε, επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων. Βεβαίως χρειάζεται επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων και εναρμόνιση σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες αλλά στην κατάσταση κρίσεων, οικονομικών κρίσεων, στις εποχές οικονομικής κρίσης χρειάζεται ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη ταχύτητα και χρειάζεται συμπίκνωση πλέον των προγραμμάτων, πιστεύω. Δηλαδή πρέπει εκείνο το οποίο είχαμε προγραμματίσει για ένα χρόνο να το κάνουμε στους 8 μήνες, ούτως ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη ένταση στην κοινωνική συνοχή και μεγαλύτερη κίνηση στην κατανάλωση. Επίσης δύο πράγματα πρέπει να δούμε οι πολιτικέ μας πρέπει να κατατείνουν σε δύο, βασικά πράγματα. Πρώτον, να καταπολεμήσουμε την ανεργία που είναι ο μεγάλος κοινωνικός κίνδυνος σήμερα και δεύτερον την ακρίβεια. Στην ακρίβεια πρέπει να δούμε και την έκδοση χαρτονομίσματος ενός ή δύο και των δύο ευρώ. Πρέπει να πάμε σε χαρτονόμισμα. Και οπωσδήποτε πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνο το πλαίσιο που να μας οδηγήσει σε αύξηση του δίκτυου εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, των ε, κυβερνήσεων αλλά και ολόκληρου της Ευρώπης ε, μεταξύ μας. Και ένα πράγμα, στον προσδιορισμό μερικών ε, φορών, επειδή μιλάμε και για το... στον προσδιορισμό του ελλείμματος θα πρέπει να βλέπουμε και μερικές ιδιαιτερότητες σε κάθε χώρα. Παραδείγματο χάρη η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα στι αμυντικέ δαπάνε. Οι αμυντικέ δαπάνε θα πρέπει να, πρέπει τις δούμε στην Ελλάδα με άλλο ο, ε, πνεύμα. Σα ευχαριστώ. Γι' αυτό έχουμε αυτή την ανταλλαγή για να μπορεί ο καθένας να παρουσιάσει τη δικιά του μαρτυρία. Τώρα για την Ιταλική αντιπροσωπεία, για το Κοινοβούλιο θα δώσω το λόγο στον Τζαν Κάρλο Τζοτζέτ ε, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμού. Ευχαριστώ. Η Ιταλία είναι και εκείνη αναγκασμένη να υποστεί τι συνέπειε τη χρηματοπιστωτική κρίση, τη οποία γνωρίζουμε το εύρο. Το τραπεζικό μας σύστημα, όπου δεν είχαμε ακόμη παρεμβάσεις επανακεφαλαιοποίησης, ε, καθώς και η χαμηλή χρέωση των Ιταλικών οικογενειών και σε σχέση με το υψηλότατο δημόσιο χρέος, που όπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε, διαθέτουμε κάποια μέτρα. Η Ιταλική κυβέρνηση διαθέτει κάποια μέσα στη, στα χέρια της, που επιτρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική, ιδιαίτερα προσεκτική, ιδίω από την άποψη τη φορολογική πολιτική. Εδώ δημιουργείται μια αντιφατική κατάσταση βεβαίω. Και αυτήν ήθελα να περιγράψω. Υπάρχει μια σοβαρή διαφορά μεταξύ του ενδεχόμενου ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τη ανεργία και τη έλλειψη νομικών μέτρων και δημοσιονομικών ε, μέσων. Ε, η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσα είναι χαμηλή και βεβαίως δεν υπάρχει και επαρκής συντονισμός. Άρα ζητάτε από τις εθνικές κυβερνήσεις, όπως ζητήθηκε συγκεκριμένα και από την Ιταλική κυβέρνηση, να κάνουν τέτοιες οικονομικές προσπάθειες ώστε να λάβουν υπόψη τους ε, και τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας. Από την άλλη όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαθέσει και τα απαραίτητα κονδύλια. Να υπογραμμίσω λοιπόν και εγώ κάποια σημεία. Πρώτον, ε, το τι συμβαίνει με τις επενδύσεις ε, για τις υποδομές, επενδύσεις εθνικές που κατά την άποψή μας θα έπρεπε να τα διαχειριζόμαστε πολύ διαφορετικά από ό,τι τώρα συμβαίνει. Και έπειτα, και σε σχέση με την παρέμβαση του Συναδέλφου, υπάρχουν και κοινωνικές συνιστώσεις πρέπει να δούμε τι γίνεται με την κοινωνική δυσφορία, τη δυσαρέσκεια που συνεχώς θα αυξάνεται και θα έχει και σοβαρές συνέπειες για τη συμπεριφορά του πληθυσμού γενικότερα υπέρ, που θα πείθεται υπέρ ή κατά του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Διότι πρέπει να παρέμβουμε και υπέρ των οικογενειών, υπέρ των πλέον πληγέντων. Ίσως ε, κάποια περισσότερα σχόλιά μου να μπορούσαν να μοιραστούν και γραπτός, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται πραγματικά χειροπιαστά μέτρα μέσω της στατικής ε, της Λισαβόνας, το Eurogroup και το ECOFIN να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο και ε, η συγχρηματοδότηση από τα Εθνικά Κοινοβούλια να προωθηθεί ως μέτρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Μπατζελή και στη συνέχεια θα έχουμε ένα νέο γύρο ερωταπαντήσεων. Κυρία Μπατζελή, στο νέο γύρο ερωτήσεων θα δώσω το λόγο στην Ισπανία στον κύριο Βίλα Χουάνα και στη συνέχεια στο Βέλγιο. Κύριε Παντζελή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέψετε δύο σύντομες παρατηρήσεις. Εάν η Ευρώπη ευθύνεται για την κρίση, θα πρέπει να έχουμε τη μεγαλοθυμία να πούμε ότι ναι ευθύνεται η Ευρώπη για, τις, ε, για την κρίση και εδώ θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν άκουσε τις παρενέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν ένα-ενάμιση χρόνο, όπου έλεγε δυναμικά για ρύθμιση και εποπτεία των αγορών αλλά η Επιτροπή με σαφές δηλώσεις αντίστοιχου και αρμόδιου επιτρόπου ανέφερε ότι οι αγορές θα ρυθμιστούν μόνο από ότι, η κρίση θα ρυθμιστεί από την αγορά. Η κρίση μας ξεπέρασε και τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα γεγονός το οποίο αν μη τι άλλο θα πρέπει να λέμε ότι είμαστε και μέτοχοι ή συμμέτοχοι σε αυτή την κρίση. Δεύτερο, για την αναδιανομή του κεφαλαίου, το reallocation όπως το χρησιμοποιήσατε, διαμέσου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Κύριε Επίτροπε, εάν πιστεύουμε ότι η αναδιανομή προς τους πολίτες γίνεται διαμέσου του τραπεζικού συστήματος πέρα ενός ιδεολογικού πιθανά ατοπήματος που ο καθένας μας έχει εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα θεωρώ ότι υπονομεύουμε το ρόλο του κράτους και δε του ρόλου του του κράτους πρόνοιας μέσα σε αυτή την κοινωνία η οποία πρέπει να είναι πάνω από αυτό απλά και μόνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο παράγει οικονομία για αυτό το είδο και δεν αναδιανέμει τον πλούτο του κράτους. Θέλω τώρα πέρα τις ε, σύντομες παρατηρήσεις θέλω να προχωρήσω σε ορισμένες σε τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, εάν στα προγράμματα εθνικής ανασυγκρότησης τα χρήματα της ρευστότητας τα οποία δίνονται στις εθνικές τράπεζες μπορούν να καλύψουν και ρευστότητα τραπεζών θυγατρικών εκτός της χώρας της οποίας είναι η βάση της τράπεζας και αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις και ποιους περιορισμούς διότι αυτό το σύστημα υποστηρίζεται από εθνικούς πόρους ενός εθνικού προπολογισμού και δεν είναι πιθανώς πρόσχημα να καλύψουμε και αδυναμίες άλλων χωρών και ρίσκα τραπεζών σε άλλες χώρες το δεύτερο ερώτημα είναι το κατά πόσον θα μπορέσουμε να συγκλίνουμε σε στοιχεία αξιοπιστία στο τραπεζό, της ε, πορείας της οικονομικής μιας χώρας όταν η Κομισιόν έχει άλλα στοιχεία, η Eurostat άλλα στοιχεία οι πιστοληπτικοί οργανισμοί άλλα στοιχεία δημιουργώντας ένα θολό τοπίο για την αξιοπιστία της κάθε οικονομίας και τέλος θέλω να επανέλθω στο θέμα του ευρωομολόγου διότι δεν είναι θέμα πότε είναι όριμη στιγμή, η στιγμή είναι τώρα διότι θα βρεθούμε με μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων μετά από δύο ή τρία χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την Ισπανία. Ο κύριος Βίλα και μετά θα έχει το λόγο το... η Βελγική αντιπροσωπεία. Eh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος ε, Αλμούνια. Βεβαίως και θα πρέπει να μιλήσει στα καταλανικά. Θα έπρεπε, θα έπρεπε, αλλά πάντως, κοιτάξτε, πρόκειται για μια γλώσσα που τη μιλάμε 10 εκατομμύρια. Άρα δεν θα πειράζει, Επίτροπε. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ 100% με τα όσα μας αναλύσατε, κύριε Επίτροπε. Θέλω τώρα ε, να, να, να κάνω κάποιε διευκρινήσει πάντω. Πρώτα-πρώτα, μα είπατε ότι πρόκειται για παγκόσμια κρίση. Άρα με παγκόσμιο τρόπο, σε παγκόσμιο οποίο θα πρέπει να επιληθεί. Όμω, είδαμε τι έγινε τώρα, είδαμε τι, τι είπαν και οι συνάδελφοι, ο σταθμό συνάδελφο από την Δανία. Κάποιε χώρε βρίσκονται σε καλύτερε συνθήκε αντιμετώπιση τη κρίση από κάτι άλλε. Υπάρχουν κάποιε σημαντικέ διαφορέ και διαφοροποιήσει που μα δυσκολεύουν όσον αφορά να αντιμετωπίσουμε αυτή την παγκόσμια κρίση. Όσον αφορά τη δική μα περίπτωση τη ε, Ισπανία, ο κλάδο των, των οικοδομών και των κατασκευών είχε πρόβλημα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σαν αποτέλεσμα σε έναν μέσο όρο ανεργίας πολύ πιο ψηλά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Φτάσουν τα 4 εκατομμύρια. Έχουμε έτσι κι αλλιώς ε, πάρα πολύ ε, μεγάλο, υψηλό δημόσιο χρέος. Φυσικά και πέρασαμε κάποια χρυσά χρόνια με πλεόνασμα στο ισοζύγιο. Όμως ακριβώς μια που θα είναι παγκόσμια η απάντηση, οι τοπικές διαφορές απαιτούν και διαφοροποιημένη κατά τόπους αντιμετώπιση όπου χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ αποφασιστική η κατάσταση αυτή γιατί θα, το, να, το, το πιο πολύ κρίσιμη κατάσταση για να γυρίσουμε σε φυσιολογική κατάσταση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά και αν δεν είχαμε κάποια ε, ρυθμισμένη οικονομία και αγορά δεν θα λειτουργούσε το σύστημα. Επομένως, το θέμα δεν είναι μόνο τι κάνουμε σε επίπεδο χρηματοοικονομικό, είναι και το θέμα του τι κάνουμε στην πραγματική οικονομία. Στις επιχειρήσεις, στις τράπεζες, τι λείπει. Λείπει το ρευστό. Άρα, δεν είναι μόνο το θέμα του να κάνουμε κάτι με παρεμβάσει στην, στα χρηματιστήρια. Γιατί πολλές φορές λαμβάνουμε εκεί κάποια μέτρα και απ' την άλλη ζορίζουμε την πραγματική οικονομία. Το 2009 επομένως ε, είναι έτος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και, και τους δύο αυτούς στόχους. Και τα ε, χρηματιστήρια και την πραγματική οικονομία που αυτή είναι η υψηλή προτεραιότητα. Δύο τελευταία σχόλια, Πρόεδρε. Χτες στο ΕΚΟΦΗΝ μιλήσανε για το έλλειμμα. Εμείς από το ΣΥΝ 2 βρεθήκαμε στο πλήν 4-5 και μιλήσανε για ένα όριο του 3, τριών μονάδων. Όμως προσοχή έχουμε τόσο πολλή ανεργία. Και προσέξτε, προτεραιότητα είναι οι άνθρωποι. 4 εκατομμύρια άνεργοι. Μεγάλο θα είναι το κόστος. Λάβετε επομένως υπό αυτό το φως αυτά τα νούμερα που αναφέρθηκαν και συμπαθάτε με για το ότι υπερεύει το χρονικό όριο. Ε, ε, Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στη συνάδελφο από το Βέλγιο. Δεν ξέρω όμως αν είστε από το, από Γερουσία ή από το Κοινοβούλιο. Ναι, είμαι από την ε, Γερουσία και είμαι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του, της Γερουσίας. Κριστιαν Η κρίση σε διεθνές επίπεδο δείχνει την ανάγκη του προληπτικού ελέγχου και ότι υπάρχουν σχετικά πάρα πολλά κενά. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της φορτής, αλλά δεν είναι και το μόνο. Στην Ευρώπη διαθέτουμε η και η ΔΕ όργανα ελέγχου, προληπτικού ελέγχου, όμως δεν υπάρχει επαρκής συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήθελα λοιπόν τη δική σας την τοποθέτηση για, την, ε, τον δεχόμενο δημιουργίας προληπτικού ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους τραπεζικούς οργανισμούς. Δεύτερη παρατήρηση, νομίζω ότι αυτό θα σταθεροποιούσε τις χρηματοπιστωτικές αγορές εάν αποσαφηνίζαμε δηλαδή την κατάσταση σχετικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έπειτα ε, στην παρούσα οικονομική κρίση οι οργανισμοί διαβάθμισης ε, παίζουν σημαντικό ρόλο γιατί εκείνοι αποστέλουν ε, ενδείξεις και σήματα προς τους επενδυτές στην Ευρώπη. Δεν έχουμε οργανισμούς διαβάθμισης, είναι όλοι αμερικανικοί, της Αμερικής μάλλον πιστεύετε εσείς για τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργηθεί ένας οργανισμός διαβάθμισης, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ένα δημόσιο όργανο, ένα δημόσιο φορέας, των 100 μελών. Ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχομαι τον ε, πρόεδρο, τον κύριο Μεστάτο, ο οποίος έκανε ιδιαίτερες προσπάθειες για να είναι μαζί μας σήμερα και να δώσω το λόγο στην κυρία Ράεβα. Έπειτα ο Επίτροπος θα απαντήσει στα ερωτήματά σας και θα κρατήσουμε τον κατάλογο των συναδέλφων που είχαν ζητήσει το ή άλλο λόγο και θα παρέμβουν αμέσως μετά, αμέσως μετά την ε, ομιλία του κυρίου Μέστατ. Μπορούμε να ενεργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγένεια και την συνεργασία σας. Κυρία Ράεβα. μπάει διορθώνει η ομιλήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε, κύριε Αλμούνια, ίσως να ήταν ενδιαφέρον για τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια να ακούσουν τις, τα σύντομα σχόλιά σα, για το γεγονός ότι οι τράπεζες που προέρχονται από παλιά κράτη-μέλη έχουν μακροχρόνια και μαζικά φαινόμενα έκθεσης στα νέα κράτη-μέλη. Οι δυσκολίε τους είναι ναι, ακόμη μεγαλύτερε σε αυτά τα κράτη, δεδομένου του σημερινού πλαισίου. Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε, θα σα δώσω τον λόγο, προσθέτοντα όμω και εγώ ένα δικό μου ερώτημα. Στο πρόγραμμα ανάκαμψη που τον έμβριο επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρχε μια ιδέα αρκετά πρωτότυπη από την άποψη των μέτρων που συνήθω ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρότεινε κάποια από τα κράτη-μέλη, εάν θέλουν να έχουν μηχανισμού παράταση ε, των μέτρων αντιμετώπιση τη ενεργεια. Γνωρίζετε πολλά κράτη-μέλη που να έχουν ενεργοποιήσει τέτοιου μέτρα. Μπορείτε να μας δώσετε μια γεωγραφική εικόνα του ποιοι τα ενεργοποίησαν και ποιοι όχι. Είναι αντός άλλω ε, ακαδημαϊκή ερώτηση και συμβολική απάντησή σας για να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα του τι έγινε και τι δεν έγινε. Ε, έπειτα μπορείτε να μας αφήσετε εφόσον το θέλετε αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας για απόψε το βράδυ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα απαντήσω σε κάποιες ε, ερωτήσεις γιατί ήδη έχουν καλυφθεί και αυτές οι ερωτήσεις ε, προηγουμένως προηγουμένως που έτσι αλλιώς μακρηγόρησα οπότε απευθείας να δούμε μερικά συγκεκριμένα σημεία πρώτον δεν συμφωνώ κύριε Μπατζηλή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται για την κρίση υποφέρει από την κρίση επλήγει από την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ούτε οι μακροοικονομικές ανισορροπίες πήγασαν από εδώ που είναι άμεσα σε αυτές οι ανισορροπίε με τις πηγές τη κρίση, ούτε από πλευρά μικροοικονομική, όσον αφορά δηλαδή την εποπτεία και η ρύθμιση των αγορών είναι η ομοιογενής η πολιτική που ακολουθείται παντού. Υπάρχουν κάποιοι φορείς που έκαναν χρηστή διαχείριση των επενδύσεων του και άλλες που δεν τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Άλλοι κάνανε καλά από τοπικές αρχές και άλλοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά του. Γιατί σε κάποιες χώρες υπάρχουν κάποιες υποπτικέ αρχές, τραπεζικές κλπ. που πάρα πολύ άσχημα τα πήγανε παρά το ότι όλοι εφαρμόζαν τις ίδιες ευρωπαϊκές διατάξεις. Εγώ είμαι υπέρ της αυστηρότερης ρύθμισης και το έχω επανειλημμένο εδώ στο Κοινοβούλιο. Και το ότι είπαμε να ξεκινήσει αυτό το, το πρόγραμμα της ε, ολοκλήρωσης των ε, υπηρεσιών πριν από 10 χρόνια είναι κάτι το οποίο οδήγησε σε 40 και πάνω πρωτοβουλίε όσον αφορά ακριβώς την, την ενοποίηση των αγορών. Οπότε και στο Συμβούλιο και, στην, και, και στο Κοινοβούλιο εμείς στείλαμε ένα σωρό προτάσεις όσον αφορά τις κεβολογικέ απαιτήσεις, όσον αφορά τους ιδίους πόρους επίσης, όσον αφορά ε, το, το, το, το, πτωχευτικό κανονισμό 2, όσον αφορά τη, του, φορεί τους φορείς αξιολόγησης και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε το φταίξιμο στην Ευρώπη. Σύμφωνοι, έπρεπε να έχουν προσπαθήσει περισσότερο, έπρεπε όλοι, όλοι να κάνουμε περισσότερο και, το Κομισιό, και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Χτες πήγα στο ΕΚΟΦΗΝ στη συνεδρίασή τους όπου είχαμε προτάσεις της Κομισιόν όσον αφορά το σχέδιο ανάκαμψης, το πώς θα εκμεταλλευτούμε 5 ε, δις ευρώ του προπολογισμού τα οποία δεν απορροφήθηκαν. Θέλουμε τώρα μα, βράχη πρόθεσμα να απορροφηθούν ούτως ώστε να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση. Και άκουσα πάνω από 6, 7, μπα, 8 ήταν οι Υπουργοί Οικονομικών από διάφορες οικονομικές χώρες οι οποίοι είπαν όχι. Όχι. Όμως η αρχή του προπολογισμού δεν είναι μόνο το Συμβούλιο, είναι και το Κοινοβούλιο. Και εγώ το ζητώ από το Κοινοβούλιο να υιοθετήσετε μια κρυστάλλινη αποφασιστική θέση κατεπηγόντως πριν το Συμβούλιο, το άτυπο της πρώτης τρίτου συνέλθει και αποφασίσει. Όμως, εάν το Κοινοβούλιο κάνει αυτό το οποίο λέμε εμείς, τότε θα τα πάμε πάρα πολύ καλά και το ζητάμε αυτό από το Κοινοβούλιο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Λοιπόν, όταν τα πηγαίνουμε καλά μας επενείται. Όταν όμως το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη δεν τα πάνε καλά, τότε να τολμήσετε να τους επικρίνετε. Να τολμήσετε. Γιατί πολλές φορές ευθύνονται τα κράτη, ευθύνονται αυτές οι υποπτικές αρχές. Δεν φταίνε πάντα. η της Κομισιόν δεν λέω ότι εσείς κάνατε αυτό το, αυτή την ανισότητα, την συμμεταχείριση, αλλά το κάνουν ορισμένοι. Επομένως υπάρχουν κάποιοι και από τους ηγέτες ακόμη σε Ευρώπη που ζητάνε περισσότερη δράση από την Κομισιόν και όταν η Κομισιόν αναλαμβάνει δράση και κατεβάζει μια πρωτοβουλία την καταψηφίζουν. Τώρα όσον αφορά τη ρευστότητα των τραπεζών για τις ε, τράπεζες και τις θηγατρικές τους σε άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουμε κάποιες αποφάσεις που εξαρτώνται από τις τράπεζες θα πρέπει να επιδέχονται από την αρμόδια αρχή κάποια υποπτία όμως επίσης υπάρχει και κάτι άλλο το, ένας άλλος ρόλος τον οποίο πρέπει να επιτελέσουν οι αρχές αυτές οι υποπτικές των χωρών όπου οι χώρες εκείνες έχουν θηγατρικές ε, υποκαταστήματα και είναι καταστημένες σε πάση περιπτώσει. Επομένως, απαιτείται σε ευρωπαϊκή κλίμακα να υπάρχει εποπτεία και έλεγχος. Και γι' αυτό χρειάζεται, ξεκινώντας από την έκθεση της ομάδας Λαροζιέρ, να πάμε σε έναν καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Και μια που έχουμε τουλάχιστον 45 τέτοιους ομίλους τραπεζικούς οι οποίοι δρούν σε ευρωπαϊκή κλίμακα, να υπάρξει σε ευρωπαϊκή κλίμακα εποπτεία. Εγώ συμφωνώ με αυτό και πρόκειται στις αμέσως επόμενες μέρες να διατυπώσουμε προτάσεις σχετικώς. Συμφωνώ και με άλλα πολλά τα οποία είπατε και τέλος η ερώτηση που αφορά τον Οργανισμό αξιολόγηση τον Ευρωπαϊκό αυτό το συζητά το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο Μητρό για να υπάρχει έλεγχος αυτών των ε, μηχανισμών αξιολόγησης, των οργανισμών αξιολόγησης. Μία από τις τρεις τέτοιες μεγάλες εταιρείες είναι εγκατεστημένη στις ΙΠΑ, η ΦΙΧΤ, αλλά βασικός της μέτοχος είναι Ευρωπαίος. Επομένως, για να μπορέσουν αυτές να λειτουργήσουν στην Ευρώπη θα πρέπει να πληρώνουν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή να γνωρίζουμε με βάση τι στοιχεία δημορφώνουν την άποψή τους. Πώς γίνεται το rating, η βαθμονόμηση, αυτή η αξιολόγηση και να ξέρουμε επίσης και τι είδους συγκρούσεις ενδεχόμενες συμφερόντων υπάρχουν τόσο ώστε έτσι να υποσκάπτεται η αξιοπιστία των συμπερασμάτων τους. Ήταν σημαντικά τα λάθη που διαπιστώθηκαν σε κάποια αξιολόγηση που κάνουν κάποιοι τέτοιοι φορείς σε κάποια προϊόντα. Δίνανε τρία αλφα σε κάποια προϊόντα που δεν τα αξίζανε. Ούτε ένα αλφα δεν έπρεπε να δώσουν. Όχι τρία που δώσανε. Τώρα, από την άλλη μεριά, πάνε να γίνουν πάρα πολύ αυστηρές αυτές οι εταιρείε και οπότε χωρίς κανένα επιχείρημα λένε για το δημόσιο χρέος. Γίνανε λοιπόν τώρα πάρα πολύ αυστηρές αυτές οι εταιρείε με κάποια, με κάποια κράτη παρά τα σοβαρά λάθη τα οποία έκαναν. Ευχαριστώ πολύ κύριε πίτροπε. Κύριε πίτροπε ευχαριστώ για όλες αυτές τις ε, ε, ε, απαντήσεις βέβαια δεν τελείωσε η συζήτηση και ο καθένας ζητά και δεύτερο πρόγραμμα στηρίξω στις τράπεζες πιστεύετε επίσης ότι θα υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες κινήσεις εν πάση περιπτώσει δεν μίλησα εγώ ούτε για δεύτερο ούτε για τρίτο πρόγραμμα για προς οποιαδήποτε κατεύθυνση όχι όχι βεβαίως απόψε θα σας ξαναδούμε ευχαριστώ και του. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος συνεδρίασής μας σήμερα το απόγευμα και θα δώσουμε τον λόγο στον ε, κύριο Φιλίπ Μεστάτ. Ξέρω ότι είχε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα ε, για πολλά θέματα τα οποία δεν είχε προβλέψει αλλά επειδή είχε δεσμευτεί απέναντί μας θέλησε να μην μας εγκαταλείψει και θα δείτε ότι είναι ε, ένας υποστηρικτής της προστιθεσμένης ευρωπαϊκής αξίας κάποια στιγμή Οπότε η συζήτηση που είχαμε απέδειξαν ότι τα προβλήματα και της προσπάθειας μονομερών λύσεων προσπαθούν να υποθάλψουν την συλλογική αντιμετώπιση την οποία πρέπει να έχουμε για την κρίση. Του δίδω λοιπόν το λόγο και μετά θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και θα ξαναπάρω τον κατάλογο των ομιλητών όπως μου είχε δοθεί. Σας υπενθυμίζω ότι θα έπρεπε ίσως να επικεντρωθείτε ε, στις μικροπιστώσεις, στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά είναι ελεύθερο και μπορείτε με οτιδήποτε να, ε, να ασχοληθείτε δεν, ε, αν έχετε άλλα θέματα που θέλετε να απευθύνετε στα Εθνικά Κοινοβούλια δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω ακριβώς όπως είπατε. Δηλαδή θα προσπαθήσω να μιλήσω για αυτό το βασικό θέμα της χρηματοδοτήσεως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μικροεπιχειρήσεων συγχρόνως διότι αφενός όταν τα πράγματα πάνε καλά διαπιστώνουμε ότι χρωστάμε πολλά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όταν τα πράγματα πάνε άσχημα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι πρώτες που πλήττονται και αυτό διαπιστώνουμε και σήμερα. Είναι λοιπόν σαφές ότι σε πολλές χώρες τα πρώτα θύματα του credit crunch όπως το ονομάζουμε είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την στενότητα δηλαδή πιστώσεων η οικονομική κρίση όπως ξέρετε ε, πλήττει 20 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καλύπτονται από τον ε, ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με κάτω από 250 απασχολουμένους είναι ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων και απασχολούν πέραν των 100 εκατομμυρίων ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ένα κεντρικό σημείο της ευρωπαϊκής οικονομίας και σήμερα διαπιστώνουμε ότι πλήττονται από την κρίση και ιδίως από το γεγονός ότι το σύστημα πιστώσεων δεν, πλέον, δεν λειτουργεί πλέον σωστά. Γι' αυτό και από πέρυσι το Σεπτέμβριο η Γαλλική Προεδρία το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών μας ζήτησαν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη χρηματοδότηση των μικρομεσών επιχειρήσεων. Όπως ξέρετε η, τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα που δημιουργήθηκε από τη συνθήκη της Ρώμης για να μπορέσει να στηρίξει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μεταξύ των οποίων και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα παραδοσιακά δανείζουμε όχι άμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί αυτό δεν είναι δυνατόν δεν μπορούμε εμείς ε, να διαπραγματευτούμε άμεσα με μία πληθώρα μικροεπιχειρήσεων αλλά εμείς δανείζουμε για να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις για να βελτιωθούν ε, να βελτιωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 5 έως 6 δισεκατομμύρια πιστώσεων διατίθενται της ίως στις τράπεζες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 2007 και το 2008 ξεκινήσαμε μία εκτενή διαβούλευση στα 27 κράτη-μέλη για να γνωρίζουμε τι ενδιαφέρον υπάρχει για αυτού του είδους το προϊόν. Ρωτήσαμε τις ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις τράπεζες βεβαίως και τους δημόσιους οργανισμούς που στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με αυτό τον τρόπο αναθεωρήσαμε και εξυγχρονίσαμε τα προϊόντα μας. Όταν λοιπόν πέρσι το Σεπτέμβριο το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών μας ζήτησαν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, είμαστε στην κατάλληλη θέση για να προσφέρουμε ένα νέο προϊόν. Νομίζω ότι ήδη θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις. Αυτό όμως που μας ζήτησε το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ ήταν να διαθέσουμε 30 δισεκατομμύρια ευρώ για να δαναδιοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 2009 ως το 2011 εκ των οποίων το ίμιση να δοθεί το 2009 και 2010 δηλαδή 15 δις και ε, έπρεπε να λειτουργήσουμε γρήγορα, πράγμα το οποίο κάναμε και ήδη κατά τη διάρκεια του 2008 μπορέσαμε να δανείσουμε 8,5 δις στις ευρωπαϊκές τράπεζες σε 16 κράτη-μέλη 8,5 δις ευρώ εκ των οποίων ε, τα, ε, τα 5 το μεγαλύτερο μέρος κατά το τελευταίο τρίμηνο διότι μας ζητήθηκε μία επιτάχυνση από το Συμβούλιο. Υπογράψαμε λοιπόν δάνεια αυτού του είδους με 16 χώρες με 75 τράπεζες με τις οποίες συνεργαστήκαμε. Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος. Καταρχήν, πλέον οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, τις πιστώσεις που τους διαθέτουμε όχι μόνο για να χρηματοδοτήσουν ε, υλικέ επενδύσεις αλλά και άλλες επενδύσεις στην έρευνα την, ε, ε, ε, την απόκτηση ενό δικτύου διανομής διαφόρων δυνατοτήτων και ένα κεφάλαιο κινήσεως working capital όταν υπάρχει μια χρηματοδότηση για λιγότερο από δύο έτη. Άρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε με αυτόν τον τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απλοποιήσαμε πάρα πολύ τις διοικητικές υποχρεώσεις των τραπεζών για απόδοση λογαριασμών για να μπορούν καλύτερα να προχωρήσουν στη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτά είναι τα δύο βασικά νέα στοιχεία. Δηλαδή ζητούμε από από την ομόλογο τράπεζά μας να δεσμευτεί γραπτός στο Συμβούλιο στο συμβόλαιο ότι ε, θα μεταφέρει ένα μεγάλο μέρος των τόκων εις ε, τις ε, επιχειρήσεις. Δηλαδή θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες χρηματοδοτήσεως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι να πλουτίνουμε τις τράπεζες και τώρα η τράπεζα ομόλογός μας θα πρέπει να δεσμευτεί σε ορισμένα θέματα ότι θα προσφέρει ιδιαίτερα προσόντα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και δεύτερον χρειάζεται διαφάνεια. Διαφάνεια προς την μικρή επιχείρηση η οποία θα πρέπει να γνωρίζει τι ωφέλη θα αποκομίσει με την επένδυση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προς εμάς διότι η ομόλογος τράπεζα θα πρέπει να μας πει σαφέστατα ποια θα είναι ε, τα ωφέλη τα οποία προσέφερε κατά αυτόν τον τρόπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα νέο προϊόν, ένα ε, σύστημα δανειοδοτήσεως ε, προς τις τράπεζες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα προχωρήσω περισσότερο σε αυτό το σημείο διότι αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δανείζουμε την τράπεζα. Δηλαδή αναλαμβάνουμε ένα κίνδυνο έναντι της τραπέζης. Πριν από δύο χρόνια θα σας έλεγα ότι αυτό δεν ε, δεν ε, επιφέρει κανέναν κίνδυνο ενώ τώρα μπορεί να υπάρξουν ορισμένοι κίνδυνοι αλλά η ενδιάμεση τράπεζα δανειοδοτεί τη μικρομεσαία επιχείρηση και αναλαμβάνει ένα μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν τον οποίο εμείς αναλαμβάνουμε προς την ε, ενδιάμεση τράπεζα. Για να μπορέσουν λοιπόν να υποκινηθούν οι τράπεζες να δανείσουν περισσότερα στις ΜΜΕ τους λέγουμε ότι αν είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις πιστώσεις ότι μπορούμε να μοιραστούμε μαζί τους τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή γίνεται μία due diligence για το σύστημα κινδύνου, αναλήψεως των κινδύνων της ε, ενδιάμεσης τράπεζας και αν μπορούμε να τις εμπιστευτούμε τους λέμε ότι αναλαμβάνουμε το ίμις του κινδύνου που αναλαμβάνουν αυτές δανείζοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θυμάστε την Βασιλεία 2, αυτό σημαίνει ότι μειώνουμε κατά το ίμιση το, το ποσό που πρέπει να δεσμεύσει η τράπεζα για να δανείσει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα μειώνονται οι κεφαλαιοχικές ανάγκες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το νέο μέσο το οποίο είναι στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι νέο και έχουμε προβλέψει επιπλέον ένα δισεκατομμύριο για ενδιάμεσα δάνεια. Δηλαδή ε, δάνεια που βρίσκονται στην ε, γκρίζα ζώνη μεταξύ το κεφάλαιο, το equity και το δάνειο, δηλαδή το χρέος. Ένα, κάτι το οποίο ονομάζουμε ε, quasi equity που ε, είναι ε, ε, μία, ένα δάνειο γέφυρα και αυτά δίδονται μέσω της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων για ύψος ενός δισεκατομμυρίου για να προωθηθούν αυτά τα δάνεια και πάντοτε το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο το οποίο έχει δύο κλάδους δραστηριοτήτων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταρχήν να δίδει κεφάλαια κινδύνου σε ειδικά ταμεία τα οποία επενδύουν προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο ε, είχε ε, διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων πέρυσι ήταν 411 ε, εκατομμύρια και εκ των οποίων για τα 300 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων διέθεσε στα venture capitals κατά τρόπον ώστε να να δοθούν εχέγγυα εις τα χαρτοφυλάκια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να υποκινήσουμε τις τράπεζες να δανειοδοτήσουν περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό γίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Τέλος, για να ολοκληρώσω τον πίνακα αυτό, θα αναφερθώ στις μικροπιστώσεις. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ε, προσφέρει εγγυήσεις για τα χαρτοφυλάκια μικροεπενδύσεων πράγμα το οποίο έχει γίνει επανειλημμένος και από την άλλη πλευρά για να σας δώσω ένα συγκεκριμένο αριθμό το, το σύνολο του χαρτοφυλακίου των μικροεπενδύσεων είναι 330 εκατομμύρια ευρώ και από την άλλη πλευρά και αυτό είναι πρόσφατο το, το ταμείο αυτό ο, διαχειρίζεται ένα, ένα ταμείο που λέγεται Jasmine και το οποίο προσφέρει τεχνική βοήθεια σε θεσμικά όργανα μικροχρηματοδοτήσεων για να εξυγχρονιστούν και χρηματοδοτεί επίσης ε, με 20 εκατομμύρια ευρώ τις συγχρηματοδοτήσεις δηλαδή για ένα ευρώ το οποίο προσφέρει ε, μία τράπεζα σε αυτά τα μικροδάνεια προσφέρουμε και εμείς άλλο ένα αυτά είναι τα μέσα τα οποία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε για να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βεβαίως δεν είναι αυτό το οποίο θα υποχρεώσει τις τράπεζες όντως να χρηματοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχω βαρεθεί να το αναφέρω διότι έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τις χρηματοδοτήσεις που δίδουμε προς τις τράπεζες 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία διαθέσαμε στις τράπεζες το 2008 τουλάχιστον το ίσο ποσό για το 2009 και πρέπει να δούμε με τι ταχύτητα οι τράπεζες όντως θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πιστώσεις για να μπορέσουν να δανειοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απλώς αυτό το οποίο λέμε σαφώς προς τους ομολόγους μας και τους εταίρους μας είναι ότι μόνο όποιος χρησιμοποιήσει γρήγορα αυτές τις νέες μορφές δανείων θα μπορέσει να υποφεληθεί στο μέλλον ε, των νέων δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Δηλαδή δεν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε τις τράπεζες, θέλουμε όντως αυτές οι πιστώσεις να χρησιμοποιηθούν για να αυξηθεί η πίστοση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί από πλευράς οικονομικής αυτό είναι το πιο βασικό και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ιδιαίτερα σαφής παρουσίαση της στράτευσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ήδη είχε ο Πρόεδρος προεξαγγείλει την πρόθεσή του για την πρόθεσή του και ιδιαίτερα την προσοχή που αποδίδουν και οι Τσέχοι συναδελφοί στο θέμα αυτό. Θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους εναλλάσσοντας Εθνικά και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βέβαια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, θα έχετε μετά την ευκαιρία να απαντήσετε στις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις. Έχω ένα κατάλογο εγγεγραμμένων για την προηγούμενη συζήτηση ήδη ομιλητών. Ίσως τώρα να μην αισθάνονται εξίσου άνετα, θα έλεγα, στο τωρινό θέμα. Πάντως, αφού έχει γίνει αυτή η αίτηση, για να λάβετε το λόγο, πρέπει να σας σεβαστώ εάν θεωρείτε ότι είναι προτιμότερο να, να μην μιλήσετε τώρα και να είστε οι πρώτοι που θα λάβετε το λόγο, το λόγο αύριο, ευχαρίστω να μεταθέσω το όνομά σα. Αλλά σα δίνω το λόγο σε κάθε περίπτωση τώρα όπω το έχουμε προβλέψει. Πρώτα λοιπόν η Πορτογαλία με τον κύριο Νίνιο Καρέιρα Περέιρα, μετά στην Ελλάδα και μετά στον κύριο Λάσλο Πέτσεκ, εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μικροπιστώσεις. Κύριε Περέιρα, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή Γεωργίας και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για την ανάκαμψη της ε, ε, ευρωπαϊκής οικονομίας Βρίσκω ανησυχητικό το να λέμε ότι η προσέγγιση μα θα είναι από πάνω προ τα κάτω μόνο και όχι το αντίστροφο. Νομίζω ότι η Ευρώπη απέτυχε τρόπον την στην κοινή πολιτική της και ιδίως ό,τι αφορά τον τομέα της παραγωγής στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες, στον ε, δευτερογενή τομέα δηλαδή, αλλά και στον πρωτογενή Επίσης, βλέπουμε πλέον η Νότια, Αμερική, η Νότια Αμερική, η Λατινική Αμερική να παράγει κάποιες φορές περισσότερο και από εμά. Και βάσει αυτή τη της αρχή, τη παραγωγική δηλαδή, να εδραιώνει την οικονομία τη. Σε ορισμένε μάλιστα απομακρυσμένες περιοχές υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην Ευρώπη των 27 πλέον κρατών μελών. Χρειάζεται λοιπόν σε ένα βαθμό ενοποίηση του πρωτογενούς τομέα και να δούμε τι συμβαίνει με τον ευάλωτο χαρακτήρα κάποιων συγκεκριμένων κλάδων στο πλαίσιο της σημερινής κρίσης. Πώς βλέπετε λοιπόν τον συσχετισμό του ανθρώπου με τον τόπο κατοικίας του, με το φυσικό του περιβάλλον και ιδίω στις λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχές, στον πρωτογενή τομέα. Γιατί κάποιες χώρες, όπως η Γερμανία, αποτελούν εξαίρεση, συνδυάζοντα τη βιομηχανία με τον πρωτογενή τομέα. Δεν συμβαίνει αυτό συνήθω στι περισσότερες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ποιε είναι οι απαρχές που χρειάζονται για την ανάπτυξη και την πραγματική πρόθεση του πρωτογενού τομέα. Ιδάλλως, δεν νομίζω να μπορεί να εδραιωθεί κανένα οικονομικό σύστημα εάν τα θεμέλια δεν τεθούν ευθύς εξ αρχής. Δεν μπορεί να συμβαίνει το αντίστροφο. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ. Υποθέτω ότι κάποιες από τις ερωτήσεις που είχαν προβληθεί για τον κύριο Αλμούνια θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν έτσι ώστε να απευθυνθούν στον κύριο τα αλλά διαφορετικά αν θέλετε μπορούμε να τις έχουμε σαν πηγή συζήτησης μεταξύ μας, αλλά για τον κύριο Μίστα δεν έχουν κανένα λόγο. Δίνω το λόγο λοιπόν στην, Ευρωπαϊ... στην ελληνική αντιπροσωπή και μετά στον κύριο Μπούτσικ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα συμφωνήσω καταρχήν με τον κύριο Φιλίπ Μεστάπ ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται πάρα πολύ. Και θα έλεγα ότι ένας από, τους λόγους που πλήττονται είναι ότι τα σχέδια διάσωσης των τραπεζών δεν, δεν εφαρμόζονται ενιαία αλλά διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Με αποτέλεσμα τα χρήματα που παίρνουν οι τράπεζες να μην περνάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην πραγματική οικονομία δεν υπάρχει δηλαδή ένα ευρωπαϊκό ταμείο για τη διάθεση της ρευστότητα και για την αντιμετώπιση της κρίσης. Δεύτερο, υπάρχει πλήρης έλλειψη αλληλεγγύης και αυτό φαίνεται από το ζήτημα που συζητούσαμε πριν από τη μη έκδοση ευρωομολόγου. Αυτή η έλλειψη θέλω να τονίσω ότι αυξάνει το κόστος του χρέους και έχει σοβαρές συνέπειες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η συνολική απώλεια για την ευρωπαϊκή οικονομία όπως την υπολόγισαν η Λόρενς Μπουν και ο, και ο Ραούλ Σόλομον της Barclays Capital ανέρχεται σήμερα σε 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι χώρες που αντιδρούν στην έκδοση ευρωομολόγων ότι η αρχή της αλληλεγγύης είναι εκείνη η οποία ενδυναμώνει την ενοποιητική προσπάθεια. Εξάλλου ανταποκρίνεται η αρχή της αλληλεγγύης και στο αίσθημα δικαίου που λέει ότι οι χώρες που αντλούν περισσότερα ωφέλη από τη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς πρέπει στην κρίσιμη στιγμή να βοηθούν τις υπόλοιπες. Ε, θέλω να ρωτήσω κυρία Πρόεδρε, είπατε κάτι στην αρχή για τη νέα αρχιτεκτονική. Μήπως στα πλαίσια της νέας αρχιτεκτονικής, εκτός από τα νομισματικά κριτήρια που υπάρχουν μέχρι σήμερα, πρέπει να δούμε για την οικοδόμηση της ενιαίας Ευρώπης και τα κριτήρια της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής στα πλαίσια ενίσχυσης του εποπτικού ρόλου που όπως είπατε πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα. Και μια δεύτερη ερώτηση. Είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις ανεξέλεκτες απολύσεις και τις αθέμητες πρακτικές που υπάρχουν στην αγορά εργασίας με όχημα ή και πρόσχημα την οικονομική κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Monsieur Κύριος πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και αν μου επιτρέπετε να ομιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την παρουσίασή του. Θα ήθελα να αφαιρθώ στα εξή θέματα. Εγώ στο ΕΛΚ είμαι πρόεδρος της ομάδας εργασίας που ονομάζεται που ασχολείται, ονομάζεται SME Circle και ασχολείται με τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα μπορούσατε λοιπόν να πείτε δύο λόγια για τις στατιστικές για την κατανομή σε επίπεδο κρατών μελών της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε ποιο βαθμό υπάρχει συνοχή στην ε, προσέγγιση αυτήν ή μήπω τα κονδύλια αυτά στρέφονται μόνο προς εκείνους που έχουν τις περισσότερες ανάγκες υπάρχει κάποια διαφορετική ε, κλίδα κατανομής Επίσης έχω την εισήγηση τη σχετική με τις μικροπιστώσεις, όπως γνωρίζετε. Ε, η έκθεσή μου ε, υιοθετήθηκε σε επίπεδο επιτροπής και θα υποβληθεί στην Ολομέλεια για έγκριση. Λέμε λοιπόν ότι οι μικροπιστώσεις στοχεύουν επιχειρηματίες που εκπροσωπούν ιδιαίτερες ομάδες εργασίας, ε, συγγνώμη, ομάδες πληθυσμού όπως γυναίκες, ε, μετανάστες, επιχειρηματίες, ε, επιχειρηματίες ε, Ρωμά, δηλαδή, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να προσφέρουν εγγυήσεις για τα δάνειά τους, αλλά είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο και να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν να τους προσφερθεί επαρκής υποστήριξη και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και από άλλες πηγές που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως λύσεις, μιμούμενοι και τις ε, ασιατικές τράπεζες. Μία λύση λοιπόν θα ήταν η, η χρηματοδότηση να προέρχεται και από μη εμπορικές τράπεζες και από άλλα ιδρύματα. Υπάρχουν διάφορα μέσα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε σαν λύσεις, δεν θέλω τώρα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν τέτοιες λύσεις. Και θα ήθελα να ερωτήσω εάν οι μικροπιστώσεις μπορούν να περιγραφούν ως κάτι διαφορετικό άλλο από αυτές οι οποίες χρηματοδοτούν επιχειρήσεις μέχρι εννέα ε, εργαζομένων. Ερωτώ λοιπόν εάν εσείς μπορείτε να βοηθήσετε εάν με κάποιο τρόπο μπορείτε να αλλάξετε τις απαιτούμενες εγγυήσεις έτσι ώστε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή φορείς αν θέλετε που δεν ανήκουν στην παραδοσιακή περιγραφή της τράπεζας να μπορούν να προσφέρουν τέτοια χρηματοδότηση. Ή αν πιστεύετε ότι είναι προτιμότερο να ε, αναλάβει το κάθε κράτος τη δική του πορεία και τις δικές του επιλογές. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ε, λάβει κάποιες πρωτοβουλίες στο πεδίο αυτό. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος στην Κυπριακή Αντιπροσωπεία τώρα και στη συνέχεια για τη Λιθουανία ο κύριος η κυρία Οντρίχη και η Κυπριακή Αντιπροσωπεία παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση που έχει κάνει ο μιλητή όσον αφορά τι ε, μικροχρηματοδοτήσει. Ε, η μέθοδο των χρηματοπιστώσεων, έχει, των μικροπιστώσεων, έχει εφαρμοστεί σε αρκετέ χώρε και κυρίω στην Αφρικανική Ήπειρο για να στηρίξει ακριβώ τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και άλλε ομάδε πληθυσμού που υπήρχαν προβλήματα και υπάρχει και σχετική έκθεση στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, στην οποία ήμουν εισηγήτρια πριν από μερικά χρόνια. Διερωτούμε, η ευρωπαϊκή επιτροπή από το 2006 έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για ανάπτυξη τη ε, μικροπίστωση και μάλιστα έχει καλέσει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία θα διευκολύνει την παροχή μικροχρηματοδότηση. Διερωτούμε ποιε χώρε έχουν ήδη προχωρήσει στην ευρωπαϊκή ένωση για να έχουν τέτοια νομοθεσία. η δική μου χώρα η κύπρο δεν έχει προχωρήσει σε ειδική νομοθεσία για μικροπιστώσει. Ε, δεν έχουμε να εγκρίνει ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο Όμω έχουμε προωθήσει με άλλου τρόπου ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη τη μικροπίστωση και πραγματικά στου προπολογισμού μα, και γνωρίζω αυτό γιατί η Επιτροπή Οικονομικών τη Βουλή παρακολουθεί στενά τα σχέδια στου προπολογισμού, υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανία και Τουρισμού που ενισχύουν την γυναικεία επιχειρηματικότητα, την νεανική επιχειρηματικότητα. Υπάρχει πρόγραμμα για το μεταποιητικό τομέα στι περιοχέ τη Υπαίθρου, σχέδιο ανταγωνιστικότητα για μικρομεσαίε και σχέδιο για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Η ερώτηση μου είναι ακριβώς επειδή είναι πολύ σημαντικό να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί στις πλήστες χώρες συμπεριλαμβανομένες και της Κύπρου αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας εάν ε, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα έχει σύντομα ε, ένα σχετικό ε, νομοσχέδιο θα θεσπίσει έναν νέο μέσο κατάλληλο για να προχωρήσει με τις μικροπιστώσεις και αν θα δώσει τεχνική βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί ακριβώς αυτός ο τομέας των μη τραπεζικών μικροπιστωτικών ιδρυμάτων στις χώρες μας. Ευχαριστώ πολύ. Λιθουανική αντιπροσωπεία. Ο κύριος Ανδρέα Ικάητης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο προσκεκλημένους μας για τις παρεμβάσεις τους. Η Λιθουανία έχει δώσει τις απαντήσεις της στο ερωτηματολόγιο που μας είχατε αποστείλει. θέλω να ρωτήσω το εξή. Και βέβαια καταλαβαίνω ότι θα είναι δύσκολο, μεγάλο έργο να συνδυάσετε τις απαντήσεις ε, όλων των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν είναι εδώ όμως ο κύριος Αλμούνια και έτσι θα ήθελα να απευθύνω σε εσά την ερώτηση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε την ανάλυση των σχεδίων ανάκαμψης, των, εθνικών σχεδίων ανάκαμψης ε, για τις εθνικές οικονομίες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις υπερβολικές ίσως γιατί αν δούμε το σχέδιο της Γαλλίας Φερρυπίν διαπιστώνουμε υπερβολικό προστατευτισμό με κίνδυνο πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την άλλη θα πρέπει να ενισχύσουμε την καλύτερη ολοκλήρωση των δημοσιονομικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ίσως και των φορολογικών και κάποια από τα ζητήματα που εμφανίζονται στην κρίση αυτή ξέρουμε πολύ καλά ότι θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν σε εθνικό επίπεδο και να επανέλθουμε στο ευρωπαϊκό για να θέσουμε τις βάσεις για μια λύση. Για τη χρηματοδότηση λοιπόν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικροπιστώσει. Είναι ένα σύστημα που ξεκίνησε το 2006. Βέβαια, εν ώψη της κρίσης επιβραδύνεται η διαδικασία. Η χρηματοδότηση των μικροπιστώσεων περνάει από τρεις τράπεζες που έχει επιλέξει το ελεγκτικό όργανο και τώρα, δεδομένης της κρίσεως, απλουστεύονται κάποιες διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε μικροπιστώσεις, κυρίως για την εκκίνηση μιας νέας επιχείρησης Και βλέπουμε ότι λειτουργεί αρκετά καλά αυτό το σχέδιο. Αλλά θα ήθελα να δω τι φρονεί ο κύριος Μίστατ ως προς το εξή, την εξή πρόταση. Θα ήταν χρήσιμο να ιδρυθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο μικροπιστώσεων στο οποίο θα συνέρεαν η τεχνογνωσία, οι ικανότητες όλων των κρατών και που θα εξασφαλιζόταν χάρη σε αυτό η υποστήριξη σε νέες επιχειρήσεις. Κυρία Φερέιρα, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά θα ακούσουμε μια τρίτη ομάδα ερωτήσεων με την γερμανική αντιπροσωπεία πρώτα και τον κύριο Λαμέλ. Κυρία Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε και πάλι μαζί μας και με και ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ακούσαμε ότι σε αυτήν την ε, φάση της κρίσης ο ευρωπαϊκός υπολογισμός είναι πολύ περιορισμένος για να αντιμετωπίσει τις ευρωπαϊκές προκλήσεις. Προκλήσεις δηλαδή ευρωπαϊκής κλίμακας. Άκουσα ότι ό,τι δεν καλύπτεται οικονομικά, ελπίζουμε θα το καλύψει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λίγο πολύ. Ότι θα παρέμβει για τις υποδομές, για την ενεργειακή πολιτική, για το περιβάλλον, για τις ε, νεοσυσταθήσεις επιχειρήσεις. Τώρα ακούμε και τα ευρωομόλογα. Αναρωτιέμαι λοιπόν σε ποιο βαθμό όλες αυτές οι λειτουργίες με τις οποίες θέλουμε να προκοδοτήσουμε τον Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κατά πόσον όλα αυτά συνάδουν με τη σημερινή του θεσμική και οικονομική διάρθρωση. Το δεύτερο μου ερώτημα έχει να κάνει με τους μηχανισμούς, τα μέσα διαχείρισης. Νομίζω ότι είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στην στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις επιδοτήσεις. Είναι δύσκολο να εγγυηθούμε ότι τις, τους ίδιους στόχους που ακολουθεί η Επενδυτική Τράπεζα Επενδύσεων τις ακολουθήσει και μια εμπορική τράπεζα. Οι οποίες ε, εμπορικές τράπεζες συγκεκριμένα τώρα αντιμετωπίζουν και έκτακτα προβλήματα. Πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λοιπόν θα πετύχει να διασφαλίσει ότι οι στόχοι στήριξης στο πλέον μικρό επίπεδο, στο πλέον χαμηλό επίπεδο των μικροπιστώσεων, πώς θα εξασφαλίσει ότι τους ίδιους στόχους θα επιδιώξουν και οι εμπορικές τράπεζες. Μια τράπεζα ιδίως που είναι γεμάτη προβλήματα και δυσκολίες για να διαχειριστεί την δική της απόφαση για να ζητήσει πίστοση. Πώς θα καταφέρει να τα φέρει εις πέρας όλα αυτά. Ευχαριστούμε και ένα τρίτο γύρο ερωτήσεων και μετά σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε στο, στο πρώτο γύρο. Στο τρίτο αυτό γύρο ο λόγος καταπόταν στον κύριο Λάμελ από τη Γερμανία και μετά στον κύριο Σχοινάρη από την Φιλανδία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι περίεργο πως ε, σήμερα ε, αναφέρουμε τέτοιους αριθμούς 3 δις, 100 ε, δις, 50 δις δεν μιλάμε για εκατομμύρια τώρα και τα χρήματα αυτά είτε προσφέρονται από τους φορολογούμενους ή αποτελούν νέα χρέη και ε, τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται θα πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικά και να αποβλέπουν σε κάποιο στόχο. Γι' αυτό η ε, τη Γερμανία είναι ένα βασικό θέμα, ιδίως η υψηλή, ε, τα υψηλά χρέη του κράτους, διότι έτσι τίθενται οι βάσεις για μια νέα οικονομική κρίση. Γι' αυτό και το ο δεύτερο πακέτο συγκυρίας θα αποφασιστεί την Παρασκευή αλλά θα πρέπει αυτό να συνάδει με μία ανώτατη ε, δανειοδότηση για την Γερμανία και τους Γερμανούς τουλάχιστον σύμφωνα με το Σύνταγμα. Ε, και το πακέτο των 100 δισεκατομμυρίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας φαίνεται σωστό αλλά τι σημαίνει ότι θα δώσει κανείς αυτές τις εγγυήσεις, ε, πώς θα γίνει η επέμβαση στην αγορά και πώς μπορεί κανείς να αποφύγει τις τρευλώσεις ανταγωνισμού. Και γι' αυτό το ίδιο ισχύει και για την οικονομική βοήθεια προς την οικονομία και την βιομηχανία, διότι με όλα αυτά τα χρήματα τα οποία μπαίνουν μέσα στην αγορά, ε, πώς είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξουν επεμβάσεις παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα μπορέσουν πλέον να αποκατασταθούν. Επίσης μας είπατε πέραν αυτής της πρώτης ερωτήσεως ότι ε, δεν μπορεί κανείς να μας υποχρεώσει να δώσουμε τα χρήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα που διαπιστώνουμε. Ότι όλες οι βοήθειες είναι καλές αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρησιμοποιηθούν αν οι τράπεζες μετά δεν τις μετακυλήσουν εις ε, τις επιχειρήσεις. Δηλαδή και οι τράπεζες τράπεζες θα πρέπει να αναλάβουν κάποιο κίνδυνο. Δεν μπορεί να τους εγγυηθεί κανείς το 100%. Θα πρέπει και αυτές να συμμετέχουν στον κίνδυνο και ελπίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες θα μείνει ένας από τους στόχους τους οποίους θα παρατηρούμε και επίσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα αποφύγουμε τον προστατευτισμό ο οποίος δημιουργείται. Ακούσαμε από διάφορους. Ο, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε ε, για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Τσεχία ε, και επίσης για τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ε, Γερμανία που είναι μια χώρα εξαγωγική. Θέλουμε να διατηρήσουμε κρατήσουμε ανοιχτές τις ε, τρίτες ε, αγορές όπως θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτή και τα γερμανική αγορά. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν στευλώσεις ανταγωνισμού μέσω αυτών των χρημάτων τα οποία θα διατεθούν στην οικονομία. Ευχαριστώ. Είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος θα σας απαντήσει. Ε, ίσως να πω και εγώ δύο αλλά παρακαλώ όποιος ενδιαφέρεται να μιλήσει, να εγγραφεί στη συζήτηση για το αργότερο όταν θα έχουμε την κυρία Νέλη Κρούς και ιδιαίτερα όταν θα συζητήσουμε για τα θέματα του, ε, της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και θα έχουμε, να, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τις αρμόδιες επιτροπής αρχές. Αντιπροσωπεία της Φιλανδίας παρακαλώ τώρα, ο κύριος Σκίνναρη και μετά η κυρία Πάιπα. Κύριε Σκίνναρη. Σκίνναρη eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής των Οικονομικών της Φιλανδικής Βουλής. Η παρέμβαση από την Γερμανία ήταν πολύ εύστοχη και ερωτώ και εγώ πώς εξασφαλίζεται ότι αυτές οι μικροπιστώσεις εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί, ότι βοηθούν αυτούς που τους έχουν ανάγκη και πώς αποφεύγεται η δημιουργία αυτό που χρήμα ελικόπτερο. Χρήμα παύλα ελικόπτερο. Πότε επίσης ερωτώ αρχίσατε να έχετε εμπιστοσύνη εσείς στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Απέδειξε στο παρελθόν ήδη ότι ήταν ιδιαίτερα απλιστό. Τώρα βλέπουμε τόσα προβλήματα πότε εξασφαλίστηκε αυτή η αίσθηση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και της τράπεζας και πώς μπορεί η Ευρώπη βέβαια να αναπτύξει πρωτοβουλίες τέτοιες, φερειπίν γύρω από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως εμείς στη Φιλανδία έχουμε κάνει έναν μέτρα γύρω από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα ή σε παγκόσμιο επίπεδο με την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενδεχομένω, αν δομή. Θα θέλαμε το ταχύτερο δυνατό να έχουμε ένα σύστημα ώστε να μην κινδυνεύουμε να πάρουν τα ενία στα χέρια τους και πάλι εκείνοι που προκάλεσαν την κρίση όταν ξαναπέσει νέο χρήμα στην αγορά. Πώς θα το εξασφαλίσετε αυτό. Πώς μετατρέπεται τώρα σε πυλώνα ηθικής και καινοτομίας ο τραπεζικός τομέας ξαφνικά. Εμείς στη Φιλανδία, όπως και είπε και ο Γερμανός συνάδελφος, ποιος τελικά θα πληρώσει το λογαριασμό. Θέλουμε όταν χορηγούνται τέτοιου είδους πιστώσεις, κονδύλια, πόροι, να ξέρουμε από ποιο προπολογισμό θα βγουν. Από τους εθνικούς, από τη φορολογία, τα λεφτά του φορολογούμενου. Η πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε και την ευκαιρία και αργότερα με τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και αύριο με την Κεντρική Τράπεζα γιατί αύριο θα έχουμε πιο πολύ τα θέματα της εποπτείας να συζητήσουμε. Η κυρία Μπάεβα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βέβαια ο Πρόεδρος Μέστα αμέσω μετά. Κύριε Μπάεβα, Πρόεδρε ευχαριστώ και αν μου, αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να μετατοπίσω κάπως την εστίαση τη συζήτηση και μια και είναι εδώ παρόν ο κύριος Μέστατ θα ήθελα να ρωτήσω τι γνώμη έχει ως προς την χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών με το, με το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Επενδύσεων και στις παρούσες συνθήκες, δεδομένου ότι εμείς στην Βουλγαρία δεν θα είχαμε υποφέρει τόσο πολύ από την κρίση εάν υπήρχε διασύνδεση από δεν θα είχαμε κυρίως από την ενεργειακή κρίση αν είχαμε τη διασύνδεση που θα μας επέτρεπε να έχουμε εναλλακτική πηγή ε, προμήθειας Φερρυπίν με τη Ρουμανία. Η Πρόεδρος, ε, είχα ήδη προαναγγείλει ότι δεν πρόκειται να ελέγξω τις ε, ερωτήσεις που θα τυπώνονταν. Θα απαντήσει ο κύριος Μέστατ πιστεύω. Και ίσως θα ήταν καλό να απαντήσετε και στις ερωτήσεις του κύριου από τη Λιθουανία για τον προστατευτισμό. Κύριε Μέστατ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Περισσότερο σε πολιτικούς ταγούς απευθύνονται και όχι στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Του του λεχθέντος βέβαια δεν μπορώ να μην ομολογήσω ότι κατανοώ βαθύτατα τα όσα είπε ο εκπροσωπός της Λιθουανίας. Ότι δηλαδή σήμερα λύση δεν μπορούμε να δώσουμε μόνο από το εθνικό επίπεδο. Και αυτό να είναι το μεγάλο δίδαγμα πιστεύω της κρίσης που διανύουμε. Ότι δηλαδή εάν θέλουμε να διαφυλάξουμε τα δημόσια κονδύλια σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, δεν μπορούμε αυτό να το πράξουμε μεμονωμένα κάθε κράτος. Αυτό ισχύει σε παγκόσμιο, γιατί η πραγματικότητα της παγκόσμιας οικονομίας είναι αυτή και ταυτόχρονα για τι μεγάλε προκλήσει του αιώνα μα, είτε πρόκειται για μια παγκόσμια επιδημία, είτε πρόκειται για την τρομοκρατία, είτε πρόκειται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, των κλιματικών αλλαγών, της φτώχειας, σε όλες αυτές τις μεγάλες προκλήσεις απάντηση μόνο με δράση συντονισμένη μπορούμε να δώσουμε, τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό επίπεδο και πάντως και στο παγκόσμιο αν υπάρχει δυνατότητα. Συμφωνώ ότι ο καθένας μόνος στη γωνιά του δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις επαρκής. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω αναφερόμενος ευρύτερα στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, διότι όντως ελοχεύει ο πειρασμό και την ανέφερε και η κυρία Φερέιρα ότι καθώ ο Ευρωπαϊκό προπολογισμό, επειδή έτσι το επιθυμούν τα κράτη-μέλη είναι περιορισμένο, ο πειρασμό είναι ότι όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα και δεν μπορούμε να το λύσουμε χορηγώντα κονδύλια από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, ο πειρασμό είναι Α ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η πρόεδρο, με συγχωρείτε, διακόπτω. Και επιπλέον σημειώνω ότι υπάρχει και ένα αρκετά δύσκολο συνομοθέτη στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή. Ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν έχει αυτόν τον περιορισμό. Ναι, αυτό μπορεί να το λέει το Συμβούλιο ω συλλογισμό, λέει ο κύριο Μέστατ. Εν πάση περιπτώσει, όταν οι δύο συνομοθέτες βρεθούν στο ίδιο μήκο κύματο, είμαι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να βρουν διαφορετικέ λύσει στα προβλήματα αυτά. Εν πάση λοιπόν, στο Συμβούλιο, σε επίπεδο Συμβουλίου, Υποπτεύομαι ότι είναι συχνό ο πειρασμό να στραφούμε προ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιατί δεν μπορούμε από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Όμω δεν είναι υποκατάσταση ένα προ ένα αυτή γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί δάνεια που πρέπει κανεί να επιστρέψει. Επιστρέφει πληρώνοντα και το σχετικό τόκο. Τόκο ίσω όχι υπερβολικό, αλλά πάντως τόκο. Άρα έχει ένα κόστος αυτή η δανειοληψία για τον ε, δανειζόμενο. Και σε πολλές περιπτώσεις μια κοινωνία, ε, μια χώρα θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιεί το μέσον της απευθείας επιδότησης, εθνικής επιδότησης από αυτό του δανεισμού για λόγους καθαρά οικονομικούς, γιατί κοστίζει. Πρώτον. Δεύτερον, δεύτερη επιφύλαξη αν θέλετε. Οι δυνατότητε δράση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων δεν είναι περιόριστε. Και γιατί. Διότι πριν χορηγήσουμε ένα δάνειο πρέπει να δανειστούμε εμείς Αντίθετα από αυτό που φαίνεται να είπε ο κύριος Λαμέλ, εμείς δεν χρησιμοποιούμε κονδύλια του προϋπολογισμού, δεν είναι χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου αυτά που διαθέτουμε. Είναι χρήματα τα οποία αναζητούμε στην παγκόσμια, στις, παγκο... στις χρηματοπιστωτικές αγορές του κόσμου. Καθημερινά και σας διαβεβαιώ ότι είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Δυσκολεύονται οι ομάδες των του προσωπικού μου να βρούνε τις λύσεις. Το Συμβούλιο μας ζήτησε να διαθέσουμε 30% περισσότερο σε δάνεια εφέτος. Πέρυσι 48 δις ευρώ διαθέσαμε σε δάνεια. Είναι ο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό με διαφορά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ξεπερνά κατά πολύ την Παγκόσμια Τράπεζα. Και μα ζητάει εφέτο το Συμβούλιο να προσθέσουμε 30%. 15 δι ευρώ δηλαδή στη δανειοδότηση αυτή. Άρα εφέτος θα πρέπει εμείς να δανειστούμε 70 δις ευρώ. Άρα είμαστε και ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειολήπτης στον κόσμο. Όταν όμω τα κράτη-μέλη μα του να δανείσουμε περισσότερα, δηλαδή να αντλήσουμε περισσότερα κονδύλια από τι αγορέ των ΗΠΑ, της Ασίας, ολόκληρου του κόσμου λίγο πολύ, από τι ίδιε αυτέ αγορέ, εμεί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ανταγωνισμό. από το Συμβούλιο, από ίδιο τα κράτη, γιατί αυτά δανείζονται πιο πολύ από εμά. Ακριβώ εκεί είναι η δυσκολία μα. Ότι δεν μπορούμε να βρούμε τη χρηματοδότηση που χρειαζόμαστε σε συνθήκες αρκετά συμφέρουσες για τον δανειζόμενο, για, αυτό, για τον πελάτη μας, αυτόν που έρθει να δανειστεί. Σας δώσω ένα παράδειγμα φρέσκο της εβδομάδας. Καλούμεθα λοιπόν να βρούμε κονδύλια γιατί μας δουν να χορηγήσουμε προς τώρα δάνεια, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για την ενέργεια και θα επανέλθω. Περισσότερα λοιπόν πρέπει να δανείσουμε και αντιμετωπίζουμε ως ανταγωνισμό. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν παράδειγμα, για 10 χρόνια δανειστήκαμε αλλά βρήκαμε μόνο δύο δις. Ενώ πέρυσι ζητούσαμε δέκα δις και τα εξασφαλίσαμε χωρίς δυσκολία. Τώρα δεν μπορέσαμε, μόνο δύο δις βρήκαμε να δανειστούμε. Γιατί, Γιατί η ισπανική κυβέρνηση, το ισπανικό κράτος, δανείστηκε εκείνο δέκα δις ταυτόχρονα με εμά και έδωσε πιο υψηλό τόκο. 90 βαθμούς βάσεως πάνω από το swap. Εμείς όμως δεν θα μπορούμε να δώσουμε τόσο. Διότι αν το κάνουμε αυτό δεν μπορούμε να προσφέρουμε συμφέρουσες συνθήκες για τον ε, μικρομεσαίο, για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι αυταπάτη λοιπόν να θεωρεί κανεί ότι μπορεί πάντοτε να κάνει περισσότερα και να προσφέρει προ τώρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αφενό μεν διότι ω εκ τη φύσεώ του είναι δάνειο και όχι επιδότηση η δική μα δράση. Πρώτον και δεύτερον διότι για να δανείσουμε θα πρέπει να δανειστούμε όχι μόνο ως προς τον όγκο και ο περιορισμός μας είναι όχι μόνο ο όγκος αλλά οι συνθήκες πάνω απ' όλα του δανεισμού που θα μας επιτρέψουν στη συνέχεια να προσφέρουμε την υπηρεσία που αποτελεί την αποστολή μας. Δανειζόμαστε και μετά δανείζουμε. Δανείζουμε τι είπα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήταν εκ των κείμενος παρεμβασής μου, θα επανέλθω. Και εδώ όντως περνούμε από έναν ενδιάμεσο, έναν μεσίτη, αυτό είναι εδώ το μέρος μόνο όμως της ε, δραστηριότητάς μας από το 40-48 δις είχαμε μόνο 8,5 με μεσητεία προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα υπόλοιπα ποσά όμως δεν τα δανείζουμε σε τράπεζες αλλά σε δημόσιες αρχές, περιφέρειες, δημοτικές αρχές, ε, κοινοφελείς υπηρεσίες ή σε μεγάλες επιχειρήσεις με τις οποίες μπορούμε να έχουμε απευθεία συναλλαγή. Αν λοιπόν περνάμε από την ε, τράπεζα ως μεσίτη, αυτό το πράττουμε για να εξυπηρετήσουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση ή μια δημοτική αρχή, γιατί δεν είναι δυνατόν εμείς να έχουμε συναλλαγή με τέτοιο μεγάλο αριθμό μικρών οφειλετών. Χρηματοδοτούμε και πέραν των τραπεζών λοιπόν. Και χρηματοδοτούμε ιδιαίτερως και τα ενεργειακά σχέδια. Και ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπάεβα για την ερώτηση της. Είναι όντως ένα ουσιαδέστατο στοιχείο και μάλιστα τώρα πια έχουμε πιστεύω συνένεση τουλάχιστον ενδιαφέρεται μια συνένεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω ότι θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να εξασφαλίσουν τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων. Απαραίτητο όμως είναι να ενισχυθούν οι διασυνθέσεις ή ε, αγωγή για τη μεταφορά της ενέργειας. Το, το είδαμε το πρόβλημα και πάλι εφέτος. Εγώ συναντήθηκα πρόσφατα με τον ε, Πρωθυπουργό της ε, Βουλγαρίας σε μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη, αφιερωμένη στον αγωγό Ναμπούκο, αλλά ταυτόχρονα μιλήσαμε και για άλλε διασυνδέσεις απαραίτητες. Στη Σλοβακία τα ίδια πράγματα συζητήθηκαν. Και Σα διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει κατά προτεραιότητα τέτοιου είδου υποδομή. Ας επανέλθω τώρα στο αντικείμενο της αρχικής μας συζήτησης, χρηματοδότηση προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικροπιστώσεις. Υπήρχαν ερωτήσεις και από τον κύριο Μπιουτσέ, ιδιαίτερα ως προς την κατανομή μεταξύ των κρατών των ποσών αυτών. Ποσόστος εμείς σαν δεν έχουμε. Αυτό είναι μια βασική αρχή στην οποία εμένουμε προαποφασιστήσα κατανομή μεταξύ των κρατών μελών δεν υφίσταται. Κάποια κρατημέλη σε τελευταία ανάλυση ενδιαφέρονται πιο πολύ η χρηματοδότηση στον ένα τομέα, ενώ κάποια άλλα σε άλλον. Εμεί μεριμνούμε έτσι ώστε συνολικά να εξασφαλίζεται μια ισορροπία, δίκαιη κατανομή, αλλά ποσόστοση κατά κράτο δεν υπάρχει. Ανακράτο μόνο δεν υπάρχει. Και αυτή η κατανομή μπορεί να ποικίλει, να διακυμαίνεται συν χρόνο. Η Γερμανία, κύριο παράδειγμα. Η Γερμανία για πολύ μεγάλο διάστημα δεν είχε δάνεια τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από την επανένωση της όμως και μετά βλέπουμε ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα ε, σχέδια που αναπτύσσονται σε περιφέρειες που έχουν καθυστέρηση την ανάπτυξή τους. Χρηματοδοτούμε λοιπόν περισσότερο σχέδια και κατά προτεραιότητα στην πρώην Ανατολική Γερμανία, τα Länder της πρώην Ανατολικής Γερμανίας και ως εκ τούτου η συμμετοχή, η αναλογία της Γερμανίας έχει ενισχυθεί. Έχει λοιπόν μεγαλύτερη εκπροσώπηση τώρα και είναι ένας από τους κύριους εποφελούμενους αν θέλετε της ε, των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά μόνο από και λόγω της επανένωσης. Δεν υπάρχουν δηλαδή ποσοστώσεις. Για τις επιχειρήσεις τώρα. Το 2008 είχαμε κατανομή σε 16 κρατημέλη. Θέλετε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, ευχαριστώ να σας προσφέρω. Αλλά πάνω απ' όλα η χώρα που επιφελήθηκε περισσότερο από τις πιστώσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν η Ιταλία. Γιατί, γιατί στην Ιταλία έχουμε από καιρό αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και με τις μεγάλες βέβαια Ιταλικές τράπεζες αλλά και σχέσεις που αναπτύσσουμε εδώ και καιρό με δίκτυο μικρότερων περιφερειακών συνεταιριστικών τραπεζών που γνωρίζουν πολύ καλύτερα το πεδίο της δραστηριοποίησής τους στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Και προσπαθούμε αντίστοιχη ε, προσέγγιση να αναπτύξουμε και σε άλλες χώρες ε, όπως την Ισπανία επί παραδείγματι όπου δανείζουμε σε ταμεία περιφερειακά, τοπικά και όχι μόνο στι μεγάλε τράπεζε. Και στα άλλα κράτη-μέλη έχουμε αντίστοιχη προσέγγιση, προσπαθώντα να προσεγγίσουμε καλύτερα τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και δανείζουμε όχι μόνο στι μεγάλε τράπεζε τη μια χώρα, αλλά και σε πιο περιορισμένη εμβέλεια τοπικέ ή περιφερειακέ τράπεζε. Κάποιε χώρε μέχρι τώρα δεν έχουν δει ουσιαστική παρουσία δική μας, Φερρυπίν, βαλτικές χώρες, μέχρι τώρα. Αν και αυτό οφείλεται ίσως σε έλλειψη ενημέρωσης Τώρα το 2009 μόλις υπογράψαμε τα πρώτα δάνεια τέτοιου τύπου με κάποιες τράπεζες στις βαλτικές χώρες. Οι χώρες του Μπένελουξ παραδοσιακά. Βέλγιο, κάτω χώρες, Λουξεμβούργο. Σουηδία, Δανία. Πρόκειται για χώρες όπου οι τράπεζες των κρατών αυτών δεν ενδιαφέρονται για δάνεια της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για δικού του λόγου και διάφορου λόγου, αλλά πάντω είναι οι χώρε που αποτελούν την εξαίρεση. Κατά τα άλλα, στι λοιπέ χώρε εκδηλώνεται ε, έντονο ενδιαφέρον για δάνεια τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυτή την εποχή. Και επανέρχομαι στι μικροπιστώσει. Προσπαθώ να εκφραστώ στο δυνατόν πιο εύγλωτα. Να σα πω το εξή. Το νέο αυτό πρόγραμμα λοιπόν, το Jasmine που ξεκινήσαμε και αναπτύξαμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συμβάλλει με 4 δι ευρώ στο πρόγραμμα αυτό. Αποσκοπούμε όχι στην εξυπηρέτηση των τραπεζών, αλλά στους θεσμούς μικροπιστώσεων, μικροχρηματοδότησης, θεσμούς που δεν είναι τράπεζες. Όμως, οι φορείς που δεν είναι τράπεζες. Αλλά ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια σε αυτού του φορεί μικροπιστώσεων, για να διευκολυνθεί η χορήγηση των μικροπιστώσεων. Και πώ το πράττουμε αυτό. Προσφέρουμε αφενό τεχνική στήριξη. Εδώ βρίσκει η χρήση η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποστηρίζουμε και τεχνικά, τεχνογνωσικά, τη μικροπίστωση, την μικρομεσαία επιχείρηση, ώστε να είναι καλύτερα σε θέση να αναπτύξει, να εξασφαλίσει την, το δάνειο που χρειάζεται, χωρίς να περνάει από την τράπεζα. Και επίσης μικροχρηματοδότηση που απευθύνεται στους φορείς αυτούς, τους μικροπιστωτικούς φορείς, αλλά σε συνεργασία με τράπεζα αυτή τη φορά. Όταν λοιπόν μια τράπεζα δεχθεί να δανείσει ένα ευρώ σε έναν μικροπιστωτικό οργανισμό, προσφέρουμε κι εμείς άλλο ένα σε δάνειο. Συμβάλλουμε. Κάποιο από τη Λιθουανία, αν δεν με ρώτησε γιατί να μην υπάρχει ένα ταμείο μικροπιστώσεων ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι θα θυμάστε σωστά. Ήταν μια αρχική ιδέα. Η αρχική ιδέα ήταν όντω να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο μικροπιστώσεων. Και είχαμε ξεκινήσει με επαφέ με διάφορου ενδιαφερομένου ενδεχομένω φορεί, διάφορου χρηματοπιστωτικού οργανισμού από τα κράτη-μέλη. Πλην όμω, αντελήφθημεν ότι. Και εδώ επανερχόμαστε στην αρχική ερώτηση το αρχικό ζήτημα καλύτερα, ότι δεν υπήρχε επαρκή αλληλεγγύη. Όλοι θέλανε να βάζουν το χέρι στον ίδιο κορβανά, αλλά θέλανε αυτό που θα προσέφεραν στον κορβανά αυτό να πήγαινε πάλι μόνο στην τράπεζα που είχε προσφέρει τα κονδύλια. Και έτσι εγκαταλείψαμε την ιδέα τη θέσπιση ενό τέτοιου ταμείου, αυτού καθ' αυτού, πλην όμω θεσπίζουμε ένα σύστημα ταχύτερο, πιο απλό, δηλαδή εφόσον χρηματοδοτεί μια τράπεζα, συμβάλλουμε κι εμείς εξίσου με τη δική μας χρηματοδότηση. Δεν εγκαταλείπω όμω την ελπίδα. Ίσως κάποια μέρα όταν πια θα έχουν ερεμήσει τα πράγματα και όταν θα έχει αποδειχθεί ότι η μικροπίστωση, η μικροχρηματοδότηση είναι χρήσιμο εργαλείο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε ότι περισσότερο τα, κράτη, τα νέα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία έχουν να διδάξουν τα παλαιότερα. Γιατί τη μικροπίστωση την έχουν αναπτύξει πολύ περισσότερο τα νέα κράτη-μέλη παρά τα παλαιά. Στα παλαιά κρατημέλη υπάρχουν αρκετέ επιφυλάξει ακόμα απέναντι στι μικροπιστώσει. Όταν λοιπόν αποδείξουμε ότι μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμο εργαλείο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε μπορούμε πιστεύω να επανέλθουμε και να ξαναεξετάσουμε την ιδέα ενός ταμείου των μικροπιστώσεων. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και εγώ ήθελα να πω τα εξή, ότι έχουμε αυτό το ερωτηματολόγιο. Αυτό το στείλαμε στα Εθνικά Κοινοβούλια και κατά κάποιο τρόπο είχαμε κάτι διαφορετικό κατά νου από ότι τα παλιότερα χρόνια. Ε, κυρίως αυτό το οποίο θέλαμε είναι να σας προκαλέσουμε ένα προβληματισμό, ε, να δούμε τι προσανατολισμό θα πάρει η συζήτηση. Δεν ζητήσαμε να, να, να, να απαντήσετε γράφο. Γιατί τρεις ε, αντιπροσωπείς αυτό κάνανε. η Λιθουανία και άλλοι δύο αυτό κάνανε σε κάποια λίγκουα φράγκα το κάνανε. Α, όπως ηλφανεί στα αγγλικά, οπότε σας έχουμε διανύμει αυτό το έγγραφο στους φακέλους που έχετε λάβει. Όμως όσοι υπέβαλαν κάποιο έγγραφο στην μετρική τους γλώσσα δεν το μεταφράσαμε και δεν το διανύμαμε. Όπως έλεγα στην αρχή, για όλους και για τον πρόεδρο Μιστάτ βεβαίω πρόκειται να προσφέρουμε μια τέτοια μελέτη από τους δικούς μας εμπειρογνώμονες μελέτη όσον αφορά ε, τα προγράμματα οικονομικής ανάκαμψης και επίσης ε, μελέτη επί των ε, προγραμμάτων υποστήριξης των τραπεζών. Το ρίσκο εδώ είναι ο προστατευτισμός και βλέπετε πόσα τέτοια προγράμματα έχουμε. Έχουμε τόσες αναλύσεις εύστοχες και πολλοί από εσά το είπανε ότι χρειάζεται να υπάρχει συντονισμός ότι να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο του προστατευτισμού κάτι που με βρίσκει σύμφωνη απολύτως. Αυτή η κρίση είναι σοβαρή. Τόσο σοβαρή που θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να κάνουμε, να καταφέρουμε το αδύνατο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα βράχη πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα και μάκρο πρόθεσμα. Κατεπήγοντα μέτρα σήμερα. Και με τέτοια κατεπήγοντα μέτρα να μπορέσουμε να δώσουμε μια καινούρια όθηση στην να δούμε τι μπορεί να γίνει με το ενεργειακό, να δούμε τι μπορεί να γίνει με το ε, κλιματολογικό πρόβλημα θα πρέπει να προσέξουμε να μην σπάσουμε τα μούτρα μας γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα ταυτόχρονα επίσης δεν μπορούμε να ζητήσουμε από κάποιον που, που, πάσχει από κάτι να γιατρευτεί μόνος δηλαδή πρόκειται για μια συλλογική ευθύνη που θα πρέπει να την ε, ασπαστούμε Όμω, δεν θα πρέπει να κοιτάει ο καθένα τα του οίκου του γιατί δεν θα τα καταφέρουμε έτσι. Και εμένα με εντυπωσιάζει αυτό το οποίο ε, ζητείται από τον πρόεδρο Ομπάμα. Αν βρεθήκαμε εκεί βρεθήκαμε σήμερα εν μέρη, όπω είπε και ο πρόεδρος ε, Αλμούνια προηγουμένω, γι' αυτό διότι ακριβώ υπάρχουν κάποιε ανισορροπίε σε παγκόσμια κλίμακα. Και πριν από δύο χρόνια είχε έρθει ο κύριο Στίγκλης και μα το είπε η πλούσια χώρα εξυπηρετεί το χρέο τη μέσω των αποταμιεύσεων των φτωχών χωρών. Όλοι επομένω λένε ότι θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να καταφέρουν οι Αμερικανοί να πετύχουν μια ανάπτυξη. Αυτό είναι σωστό, αλλά όμως δεν πρέπει να γίνει με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί. Θα πρέπει αυτή η όθηση στην οικονομία να γίνει με τρόπο ευφυή και να μην ε, αγνοήσουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Να μην έχουμε ζυζάνια προστατευτισμού. Να γίνει μεταρρύθμιση, να γίνει αναθεώρηση των οικονομικών μοντέλων που χρησιμοποιήσαμε τα τελευταία πολλά χρόνια. Πολύ σημαντικό. Και τώρα σας λέω την προσωπική μου άποψη, δεν σας μιλώ σαν πρόεδρος. Αν ρίξουμε μια ματιά στο τι γίνεται στη ΣΥΠΑ, έχουμε μια αλλαγή του πρότυπου. Τώρα πάμε προς καλύτερη αναδιανομή του εισοδήματος. Να είναι πιο βιώσιμο ο πλευρά ενεργειακής, από πλευρά περιβαλλοντική στο οικονομικό μοντέλο. Να είναι καλύτερο από το σημερινό όσον αφορά τώρα την Κίνα. Πάμε προ ανάπτυξη εσωτερική αγορά για να σταματήσει η Κίνα να είναι ένα εργαστήρι που εξάγει. Εξάγει σε εμά υπό τις συνθήκες αυτές που δεν είναι οι μας επιχειρήσεις. Άρα θα πρέπει ταυτόχρονα να κάνουμε πολιτική μακροπρόθεσμη, βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη. Να μην πούμε εγώ σήμερα θα κάνω αυτό και όποιος με, με διαδεχθεί στις επόμενες εκλογές μα, ξέρουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει το, το έργο που ξεκινήσαμε εμείς. Άρα χρειάζεται παράλληλα να προχωράμε σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο όσοι θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό και ότι θα πρέπει έτσι να βρεθεί η λύση εάν δεν το σκεφτείτε αυτό τότε δεν θα καταφέρετε τίποτα Αναλαμβάνω τι ευθύνε μας το είπε και η ο Λούλινγκ από το Λουξεμβούργο τρομερό γιατί σήμερα έχουμε μια νομοθεσία χωρίς αρχιτέκτορα η αρχιτεκτονική ποια θα είναι τι θα γίνει αύριο, πώ θα γίνεται η εποπτεία παγκόσμια, η πανευρωπαϊκά, δεν ξέρω, κανεί δεν ξέρει, οπότε και εμεί κάθε μέρα προσπαθούμε να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι το θεμέλιο τη Ένωση το είπε και ο Επίτροπο Αλμούνια. Η εσωτερική αγορά, ο ανταγωνισμό, αυτό που έχουμε οικοδομήσει τόσα χρόνια, όλα αυτά τίθενται να αμφιβόλω και θα έχουν κακή κατάληξη. Κάτι το οποίο το θέλει κανείς. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι τόσο σημαντικό να ε, καταπολεμήσουμε τον προστατευτισμό να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε αυτούς που χτυπήθηκαν από την κρίση παρασύρθηκα δεν γίνεται αλλιώ. αλλά θα ήθελα και εγώ να σας πω τις δικές μου απόψεις πάνω στις ερωτήσεις σας τώρα για έναν τελευταίο γύρο ερωτήσεων, ε, να δούμε ποιοι έχουν ζητήσει ήδη το λόγο, να δούμε μην ξεχάσουμε κανένα και κατόπιν να δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο Μέιστατ. Από τις κάτω χώρες έχει ζητηθεί ο λόγος τώρα. Ο κύριος Μπαλτασάρ από την Ολλανδική Γερουσία. Και κατόπιν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κυρία Φαντενμπουργκ. Θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Από την Αυστρία, ζητείτε το λόγο. Δύο. Πρώτα πρώτα, Ολλανδία. Πίτερ Ρόμσχερτ ονομάζομαι βουλευτής στους χριστιανοδημοκράτες στη χώρα μου. Δύο παρατηρήσεις έχω να σας υποβάλω. Πρώτα πρώτα ότι όλοι έχουμε τόσο μεγάλο χρέος αυτό το 3% είναι ένα όνειρο, όνειρο απατηλό. Πώς θα εξασφαλίσουμε το ότι δεν θα πάρουμε τον δρόμο της αστάθειας Για μην καταλήξουμε δηλαδή κάπου όπως η Ισλανδία. Τους κορυδεύουμε τώρα, αλλά εάν βρεθούμε σε μια βαθιά ύφεση και έχουμε φτάσει σε καταστάσεις μεγάλων ελλημάτων όπως προαναφέρατε, τι θα κάνετε άμα θέλει η Γαλλία και η Ισπανία δέκα δις την ίδια μέρα, πώς θα βγούμε το διέξοδο. Δεύτερη ερώτηση αφορά την τράπεζα επενδύσεων. Θεωρείτε ότι θα μπορέσει κάτι να κάνει γιατί λέμε για να δεις έξτρα κεφάλαιο για τις τράπεζες μα αυτό δεν είναι τίποτα γιατί οι Γερμανίες για τι δικές του τράπεζες και τράπεζες χρησιμοποιούν 480 δις άρα τι μπορεί να βάλει παραπάνω η ΕΤΕ, πού θα τα βάλει σε σχέση με τις εσωτερικές πολιτικές που χρησιμοποιούν τέτοια τεράστια ποσά σε Γερμανία, στην Αγγλία και στην Ολλανδία, τη χώρα μου. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Τώρα ο Γιος Μπαλτασάρη από την Ιταλική Γερουσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε για αυτό το έγγραφο της δικής μας γερουσίας για την χρηματοοικονομική κρίση. Είναι συνθετική δουλειά. Τρεις μήνες δουλέψαμε. Και ακριβώ κρίθηκε πάρα πολύ σωστό το να σε όλου. Επίσης ευχαριστούμε και τον Πρόεδρο Μάιστα διότι μας ανέφερε μας και είπε ότι και εμείς είμαστε ένα παράδειγμα προς μίμηση για τις ΜΜΕ όσον αφορά αυτές τι επενδύσει τη ΕΤΕ και άμεσα να χρηματοδοτήσει τις τοπικέ τράπεζε. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να σταθεί κοντά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην πράξη επιτόπου, διότι ακριβώς το ποσοστό των πιστώσεων που απευθύνεται αυτές, σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σαφώς ανεπαρκές και δυσανάλογο σε σχέση με αυτό που απευθύνεται στις μεγάλες. Ε, πρόεδρε, πάντως έχουμε και έναν φόβο, διότι αν οι πόροι των κρατών κατεξοχήν κατευθύνονται όπως έχει, έχει γίνει συνήθεια να συμβαίνει Είπατε κι εσείς Επιτροπέ ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια ότι τα κονδύλια που διατέθηκαν έφταναν στο 2-3% του ΕΕΠ, αλλά συνολικά τα κονδύλια που θα στηρίξουν τα χρέη των μεγάλων τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα κονδύλια που θα απευθυνθούν στις οικογένειες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναλογικά τουλάχιστον. Άρα ο φόβος μας τελικά είναι ο εξής, αν τα δημόσια κονδύλια ή εκείνα που θα μπορούσε να προσθέσει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε μεγάλο βαθμό στηρίζουν μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλες τράπεζες και μεγάλες εταιρείε. Ο κίνδυνος δεν είναι μετά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πληρώσουν ε, διπλά τις συνέπειες της κρίσης αυτής. Από τη μια από την άποψη των πιστώσεων και από την άλλη των τιμών, δηλαδή των επιτοκίων. Σας θέτω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Πρόεδρε, ζούμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο παράδοξο που ίσως να μας αναγκάσει να επινοήσουμε και νέες οικονομικές θεωρίες. Από τη μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φροντίζει για τη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, κινδυνεύοντας επίσης να φτάσουμε και σε μια παγίδα της ρευστότητας, τη λεγόμενη liquidity trap. Από την άλλη όμως το τραπεζικό σύστημα έχει μπλοκαριστεί γιατί δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη μεταξύ των τραπεζών. Υπάρχει λοιπόν η δυσκολία με την ε, παγίδα αυτή της ρευστότητα, αλλά υπάρχει και αυτή η κάμψη της πραγματικής οικονομίας. Ένα πραγματικό crunch που αντιτίθεται στην τραπ. Είναι λοιπόν πραγματικά επικίνδυνο όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα μπορούσαν να φανταστούν τουλάχιστον για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να προβλέψουν εγγύηση για το διατραπεζικό σύστημα ώστε η ρευστότητα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπορέσει να περάσει και στο παραγωγικό σύστημα. Και έπειτα, τι άποψη για τη γαλλική απόφαση να προβλεφθεί κάτι σαν ένας ε, αστικός ε, ελεγκτής για τις μικροπιστώσεις, διαμεσολαβητής, για τις πιστώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάποιος που να χρησιμεύει δηλαδή ως ενδιάμεσος, να ελέγχει τους όρους, τις ποσότητες και τις τιμές με τις οποίες φτάνουν οι μικροπιστώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ίκε Βάγκεμπουργκ και μετά η Αυστριακή αντιπροσωπή και θα έχουμε ολοκληρώσει με τους ομιλητές για σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που δεν άκουσα την εισαγωγή σας, γιατί ε, πάντοτε παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τα σχόλιά σας. Άκουσα όμως ε, πώς απαντήσατε σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά ε, με την ε, ε, χρηματαγορά όπου ε, υπάρχουν πάρα πολλά ομόλογα κρατικά από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα σχολεία σας σχετικά με το θέμα αυτό. Αντιλαμβάνουμε ότι προσπαθείτε κάπως να συντονίσετε αυτά τα κράτη-μέλη. Δεν θα ήταν όμως ευκαιρία να προχωρήσετε πολύ περισσότερο και όχι απλώς να συντονίσετε αυτά τα θέματα των ομολόγων και αντί να προσπαθήσετε να τα συγκεντρώσετε, να βρείτε ε, κάποιο πιο, ε, κάποια άλλη δραστηριότητα πιο επικερδή και πιο αποδοτική ε, και πιο φθηνή σε τη διεθνή χρηματαγορά διότι βλέπουμε τα ομολογιακά τα, τα ομοσπονδιακά ομόλογα στις Ηνωμένε Πολιτείες. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε από την πείρα σας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως ενδεχομένως όχι τώρα αμέσω, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να μας δώσετε ε, ε, κάποιους αριθμούς σχετικά με τα προσόντα, ε, τα κέρδη και τις οικονομίες που θα κάνουν τα κράτη-μέλη εάν προτιμήσουν την τράπεζά σας για να εκδώσουν από κοινού ομόλογα. Ευχαριστώ. Η Αυστριακή Αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σχετικά με τις μικροπιστώσεις έχω μία διαπίστωση έχουμε διάφορες τράπεζες στην Αυστρία που χορηγούν μικροπιστώσεις πάντοτε όμως υπάρχουν προβλήματα διότι το διοικητικό κόστος και η επιτήρηση είναι μέτρα τα οποία ε, δίνουν την ευκαιρία στις τράπεζες να μην δίνουν Τέτοιε τέτοιες μικροπιστώσεις και να τις αρνούνται. Έχω και μία γενική παρατήρηση. Ε, τι νόημα έχει εάν στα ευρωπαϊκά κράτη χρησιμοποιούμε τόσο αυστηρά τη συνθήκη Βασιλίσσιας Δία τη στιγμή που στις Ηνωμένε Πολιτείες αγνοείται τελείως ε, το, η συνθήκη αυτή. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Mm. Καταρχήν σχετικά με συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ιδίως ε, του ε, βουλευτή από την Ολλανδία που είπε ότι αυτό το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε στις τράπεζες είναι σχετικά λίγο σε σχέση με ε, τα, το ότι προσέφεραν τα κράτη για να σώσουν το τραπεζικό σύστημα. Αλλά η δικιά μας παρέμβαση είναι κάπως διαφορετικής μορφής. Δηλαδή ο στόχος μας δεν είναι να βοηθήσουμε τις τράπεζες ε, εκεί που στοχεύουμε εμείς είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την παροχή πιστώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δανείσουμε φέτος στις τράπεζες είναι λίγα σε σχέση με ό,τι έχουν προσφέρει τα διάφορα κράτη. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξού και οι όροι τους οποίους περιλαμβάνουμε στις συμβάσεις δανειοδοτήσεως για τις ενδιάμεσες τράπεζες, δηλαδή πρέπει να μεταφέρουν ε, κάποιο προτέρημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταρχήν από πλευράς ε, όγκου. Για κάθε ευρώ που δίνουμε εμείς στην τράπεζα πρέπει να αποδείξει ότι αυτή έχει χορηγήσει 2 ευρώ δάνειο στην μικρομεσαία επιχείρηση. Θα πρέπει δηλαδή να αποδείξουν ότι Εάν δώσουμε 250 εκατομμύρια ευρώ θα έχουν δοθεί 500 εκατομμύρια ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή να αποτελέσουμε ένα μοχλό για να, αυξηθούν, να αυξηθεί η δανειοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στα νέα συμβόλαια τα οποία διαπραγματευόμαστε τώρα επιβάλλουμε και την υποχρέωση να μεταφερθεί με ένα ελάχιστο χρηματικό προσόν. Δηλαδή θα πρέπει τουλάχιστον τουλάχιστον ένα ελάχιστο ποσοστό αν το επιτρέψει η αγορά γιατί οι συμβάσεις που υπογράφουμε τώρα προβλέπεται ε, τουλάχιστον να υπάρχει μία διαφοροποίηση επιτοκίου ε, των 0,45 ε, points για να μπορέσουμε ίσως από πλευράς όγκου να κάνουμε κάτι μικρό αλλά πιστεύουμε ότι συσσωρευτικά, αθρηστικά όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν τον όγκο των πιστώσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρακολουθούμε δε με τι ρυθμό οι τράπεζες οι οποίες χρησιμοποιούν τις πιστώσεις αυτές τις χρησιμοποιούν για να χρηματοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε τώρα την κατάσταση διαφορά ρετικά μεταξύ κρατών. Άλλα κράτη τις χρησιμοποιούν πολύ πιο γρήγορα και άλλα πολύ πιο αργά. Γι' αυτό και θέλουμε να συνεχίσουμε την πίεση κατά τρόπον ώστε να χρησιμοποιηθούν όντως οι πιστώσεις αυτές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στις συμβάσεις τις οποίες υπογράφουμε τις τράπεζες έχουμε το δικαίωμα να στείλουμε δικούς μας εσωτερικούς ελεγχθές για να δούμε πώς το σύστημα εφαρμόζεται. Όσον αφορά την ανησυχία που εξέφρασε ο εκπρόσωπος της ε, Ιταλικής Γερουσίας. Ε, τον ευχαριστώ που μας είπε ότι στην Ιταλία προσπαθήσαμε να διαφοροποιηθούμε. Είπε ότι η εμπειρία ήταν θετική και αυτή είναι και δικιά μας άποψη και γι' αυτό τώρα προσπαθούμε και σε άλλα κράτη-μέλη να ε, κάνουμε τέτοιες συμβάσεις δανειακές με περισσότερες ενδιάμεσες τράπεζες ενδεχομένως συνεταιριστικές κρατικές ή περιφερειακές ε, τράπεζες, ε, ταμιευτήρια, τα οποία ε, πρόσκυνται περισσότερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά έναν διαμεσολαβητή για τις πιστώσεις, μου ρωτήσα τη γνώμη μου. Βεβαίω υπάρχει σε ορισμένε χώρε. δηλαδή παραδείγματο χάρη στο Βέλγιο εδώ και πολλά χρόνια. Εάν μία μικρή τράπεζα αρνηθεί να χορηγήσει μία ε, ένα δάνειο και ε, διαφωνήσει η ε, μικρή επιχείρηση μπορεί να προσφύγει σε έναν διαμεσολαβητή και να ζητήσει τους λόγους της αρνήσεως. Στην κυρία Βαντενμπύρτ θα πω ότι το σχόλιο της είναι λογικό. Και ξέρετε ότι αυτό το πρεσβεύουν ορισμένοι και ιδίω ο Ζων Κλοντ Ιούνκερ, ο πρόεδρος του Ευρωγκρουπ και Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, ο οποίος ε, είπε να υπάρξει ένα τέτοιο πουλ, ένα σύνολο το οποίο θα επιτρέψει να δοθούν ε, δάνεια με καλύτερους όρους, διότι αυτή τη στιγμή εμείς ε, δανειζόμαστε με καλύτερα επιτόκια από ότι ορισμένοι από τα μέλη μας, η μετοχή μας, δηλαδή τα κράτη-μέλη. Διότι όλοι, όλα τα κράτη είναι μετοχή, υπάρχει ένας μέσος όρος μεταξύ των κρατών, άρα εμείς μπορούμε να δανειοδοτηθούμε με καλύτερες, καλύτερους όρους και γι' αυτό ε, ε, ίσως γνωρίζετε ότι η ιδέα αυτή έχει απορριφθεί από συναδέλφους του Jean-Claude Juncker στο Eurogroup αλλά το επιχείρημα ήταν ότι αυτό θα φερούσε ε, ένα κίνητρο για τη δημοσιονομική πειθαρχία και αυτό που είπαν οι αντίθετοι προς την, αυτή, ε, προς ιδέα αυτή θα ήταν ότι θα πρημοδοτούσε κανείς αυτούς που τους ξέφυγε το δημόσιο έλλειμμα και θα τους πρημοδοτούσαμε. Και γι' αυτό εν ονόματι της διατηρήσεως της ε, δημοσιονομικής πειθαρχίας έχουν απορρίψει αυτή τη λύση. Και αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση του ε, Ολλανδού βουλευτού, διότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πώς θα υπάρξει δημοσιονομική ισορροπία μεσοπρόθεσμα, διότι είτε το θέλουμε είτε όχι, ορισμένες προκλήσεις θα συνεχίσουν να υφίστανται και ιδίω η δημογραφική γύρανση. Δεν θα γίνουμε όλοι πιο νέοι επειδή υπάρχει μία οικονομική κρίση, άρα οι επιπτώσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις εθνικ... τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Εάν λοιπόν δεν ισοσκελίσουμε το προπολογισμό μας σύντομα θα είμαστε σε μερικά χρόνια σε δινή θέση. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει από αυτές τις συνθήκες να υπάρξουν προγράμματα ανακάμψεως και μέσω της δημοσιονομικής οδού. Εγώ ήμουν πολύ επιφυλακτικός μέχρι τώρα, διότι προέρχομαι από μια χώρα που χρόνια μας, μας ξέφυγε ο προπολογισμό και ε, ήμουν υπουργό Οικονομικών και μια φορά είχαμε έλλειμμα προπολογισμού 13% και χρειάστηκε να λάβουμε μια ολόκληρη σειρά από αντιλαϊκά μέτρα. Λοιπόν, ε, θέλω να πω ότι υπό τις ισχύουσες συνθήκες επειδή υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την ε, ανάκαμψη και δεν υφίστανται σήμερα ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή είναι ε, ανάκαμψη δια της δημοσιονομικής οδού αλλά ισορροπημένη με συγκεκριμένα μέτρα διότι φοβάμαι ότι για την δημοσιονομική ανάκαμψη θα δικαιολογήσει κανείς δαπάνες που δεν έχουν καμία σχέση και θα επιτρέψουν απλώς να δώσει κανείς προεκλογικά δωράκια. Χρειάζεται λοιπόν εστιασμένη πολιτική ε, και μέτρα ορισμένης διαρκείας, δηλαδή για δύο χρόνια και τέρμα στο τέλος του 2010. Τα μέτρα αυτά θα πάψουν να ισχύουν στο τέλος του 2010 εκτός αν αποτιμήσουμε ότι πρέπει να συνεχιστούν. Πρέπει πρέπει πάντοτε όμως να μας απασχολεί το θέμα ότι πρέπει να επανέλθουμε στην δημοσιονομική ισορροπία ε, σύντομα, διαφορετικά θα έχουμε ένα ζωφερό μέλλον. Ευχαριστώ τον ε, Πρόεδρο για αυτά τα πολύ σημαντικά σχόλια και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο ή στον συνάδελφο Γιάν Χάτσα για να, για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος των συζητήσεών μας και μετά θα σας δώσω συγκεκριμένες ε, ε, ε, οδηγίες για το τι μέλη γενέστε μετά τη συνεδρίαση αυτή. Σας δίνω το λόγο συνάδελφε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Όσον αφορά αυτό το πρώτο μέρος της συζητήσεώς μας είναι πάρα πολύ θετικό το ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικές είναι οι ΜΜΕ για τις οικονομίες των κρατών μελών και για την απασχόληση ε, το ίδιο ισχύει και για την ε, Προεδρία μου Ακριβώς εκεί θέσετε στην προσοχή μας το πώς θα έχουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία και θα εφαρμόσουμε σας ε, προείπα για την θέσπιση του νόμου των ΜΜΕ και το πρόγραμμα δράσης και θα συνεχίσουμε με τέτοια διαδικασία νομοπαρασκευαστική όσον αφορά τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ αλλά και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία. Επίσης θα ασχοληθούμε με κάποιες υπερημερίες πληρωμών και θα ξεκινήσουμε από τον Μάρτιο του 2009. Θα συμμετάσχουμε όσο γίνεται πιο δυναμικά στην εβδομάδα για τις ΜΜΕ. Σκοπός αυτής της εκδήλωσης θα είναι ότι θέλουμε να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο για το τι ισχύει σε κάθε επίπεδο. Να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να αρχίσει να δημιουργεί επιχειρήσεις τέτοιες. χρηματοδοτική κρίση και οι λύσεις. Θα συνεχίσουμε την συζήτηση αύριο που θα έρθει και ο Υπουργός κ. Κάλουσεκ. Αυτό θα είναι το θέμα μας. Προς το παρόν, αρκεί να σας ευχαριστήσω εσάς, την ε, Οικονομική Επιτροπή, σας ευχαριστώ για την τόσο ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι πάντα κάτι ευχάριστο και τα συμπεράσματα είναι πολύ χρήσιμα. Θα αντιλήσουμε συμπεράσματα από αυτά που είπατε εσείς, ότι δηλαδή θα πρέπει από κοινού να βρούμε λύση αυτά τα προβλήματα, γιατί το πρόβλημα μας αφορά όλους στην Ευρώπη και έτσι θα πρέπει να προσεγγίσουμε και την λύση αυτού του προβλήματος. Αγαπητέ συμπρόεδρε, κανείς δεν θα μπορούσε να τα διατυπώσει καλύτερα όσον αυτά τα συμπεράσματα, γιατί ακριβώς θα πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις να πάρουν το μήνυμα ότι δηλαδή η διέξοδος θα ανεβρεθεί μόνο αν προχωρήσουν προς αυτήν όλοι μαζί. Εδώ. Τώρα να διακόψουμε τις εργασίες μας και να δώσουμε ραντεβού στις 7.30. Στο Ισόγειο, στην τραπεζαρία, απέναντι. Και κατόπιν να φάμε, να συζητήσουμε, αλλά όχι και παραβολή, ούτως ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν όσοι θέλουν και κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε πιο, πιο στενές επαφές όλοι μαζί.